Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... seats. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Καθίστε, παρακαλώ. Plenty of, of seats. Έχει θέσεις εδώ. I hope that the other members will... Ελπίζω να έρθουν και οι υπόλοιποι λίγο αργότερα. Πάντα 9 η ώρα το πρωί πρόβλημα είναι, αλλά παρόλα αυτά να ευχαριστήσω όλους εκείνους που είναι ήδη εδώ και να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία θα γίνει σήμερα το πρωί και το απόγευμα και αύριο το πρωί. Έχετε δει την ημερησία διάταξη, σας έχει διανεμηθεί. Μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο μερίσας διάταξης ε, για τη συνεδρίαση σήμερα και αύριο. Υπάρχει κάποια πρόταση. Όχι, επομένως εγκρίνεται η μερίσα διάταξη. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων από τις 18 ε, Μαΐου και τις συνεδρίες 29 και 30 Μαΐου του 2017. Το σχέδιο πρακτικών είναι διαθέσιμο ε, στο διαδίκτυο, όπως γνωρίζετε, προτείνω ως συνήθως, εάν δεν υπάρξουν ε, ενστάσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται οι, ε, τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Δεν βλέπω σχόλια και προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο, ανακοινώσεις της Προέδρου. Επιτρέψτε μου να σας κάνω τρεις ανακοινώσεις μόνον για να σας υπενθυμίσω τι συνέβη μεταξύ των δύο συνεδριάσεων δηλαδή. Να ξεκινήσω από χθες. Είχαμε τη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επίπεδου για την απλούστευση ε, στο κτίριο Μπερλεμόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήμουν προσκεκλημένη. Ε, για την ε, ε, κατά πάσα πιθανότητα τελευταία επίσημη συνεδρίαση αυτής της ομάδας υψηλού επίπεδου εκ μέρους της Επιτροπής Ρέτζη. Η συζήτηση αφορούσε τις τελικές συστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν από την ομάδα υψηλού επίπεδου και έχουν διανεμηθεί και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη. Η παρέμβασή μου στάθηκε στο ρόλο της διαδικασίας απλούστευσης, ε, ενημέρωσα την ομάδα υψηλού επίπεδου και όλους τους ενδιαφερομένους και τους ε, επιτρόπους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση για τις ε, δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι εμείς ε, ασχολούμαστε με τα θέματα της απλούστευσης με πολύ δραστήριο τρόπο. Κάναμε ανταλλαγή απόψεων δύο φορές με τον πρόεδρο της ομάδας υψηλού επίπεδου. Έγινε και σχετικό ειδικό εργαστήριο και συμπεριλάβαμε και την απλούστευση σε κάθε μία από τις εκθέσεις που εγκρίναμε εδώ στο Κοινοβούλιο τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε λοιπόν δραστήριοι εταίροι ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της απλούστευσης και το μόνο θέμα το οποίο ετέθη στη διάρκεια αυτής της συζήτησης ήταν τι θα γίνει με το φάκελο Omnibus. Ε, εμείς ε, έχουμε ήδη γνωμοδοτήσει εδώ και δύο μήνες. Ε, ελπίζω να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος ε, το Σεπτέμβριο και ελπίζω ότι η νέα Εσθονική Προεδρία θα ε, φροντίσει να οργανώσει αυτούς τους τριμερείς διαλόγους. Ε, είχαμε παρουσία δύο επιτρόπων στη συνεδρίαση. Ήταν εκεί η Επίτροπος Κρέτσου, που είναι αυτή η οποία άλλωστε ε, ξεκίνησε και αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου, και η Επίτροπος Τάισεν. Ε, και οι δύο αναφέρθηκαν ε, στο πολύ σημαντικό ρόλο της απλούστευσης των κανόνων και για την παρούσα περίοδο αλλά και για τη μελλοντική περίοδο μετά το 2020 δηλαδή. Αυτά λοιπόν τα της ομάδας υψηλού επίπεδου. Οι συστάσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ε, και όπως ε, είπε και ε, κάποιος συνάδελφος ίσως είναι λίγο πολύ δικητικές, αλλά υπάρχει η αίσθηση της ανάγκης της απλούστευσης. Η δεύτερη ανακοίνωσή μου αφορά την κοινή συνεδρίαση Ρέτζι ε, Κοτέρ ε, για την ε, εταιρική σχέση για το αστικό θεματολόγιο που έγινε στις 29 Ιουνίου. Κάποια από τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Ήταν παρούσα και όλη η Επιτροπή Κοτέρ στη διάρκεια αυτής της ακρόασης. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις δραστηριότητες των εταιρικών συμπράξεων, αλλά και ε, πώς μπορούμε μέσω αυτών των συμπράξεων να εμπλέξουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες ε, στη συζήτηση για το ρόλο των Ευρωπαϊκών Πόλεων, να ενημερώσουμε τους πολίτες για τους στόχους μας και τα επιτεύγματά μας και επίσης ε, Συζητήθηκε και πώς μπορούμε να έχουμε συμμετοχή και διαφόρων ομάδων της κοινωνίας ε, ε, στα δημοτικά συμβούλια, αλλά και να έχουμε και συμμετοχή επιχειρήσεων και άλλων οργανώσεων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις και νομίζω ότι είναι διαθέσιμες αν σας ενδιαφέρουν. Τρίτη ανακοίνωση. Ε, το Φόρουμ της Συνοχής, το οποίο διεξήχθη στις 26 και 27 Ιουνίου και η Επιτροπή μας είχε μεγάλη εκπροσώπηση στη διάρκεια των συζητήσεων. τόσο στη συζήτηση εν γέννη, αλλά είχαμε και τρεις ε, εξημών που ήταν αρμόδιοι για τα πάνελ. Ο, η κυρία Κρέλ, ο κύριος Φανίστερλο και εγώ ήμασταν πρόεδροι τριών εργαστηρίων. Η κυρία Βέστφελ συμμετείχε ενεργά και αυτή στις συζητήσεις. Ε, Υπήρχε λοιπόν πολύ καλή εκπροσώπηση σε αυτό το φόρουμ συνοχής ε, και η μόνη παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω για εκείνους που δεν είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε ιδιαίτερα ενεργά στο φόρουμ. Ε, δηλαδή το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήρθε και ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οι περισσότεροι επίτροποι συμμετείχαν στην ε, Ολομέλεια με τις, ε, και με βασικές ομιλίες, αλλά συμμετείχαν και στα εργαστήρια ε, με κέρυες ομιλίες. Το φόρουμ ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τίποτα πολύ εντυπωσιακό βέβαια αλλά ε, ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ενδιαφερομένους και να παρουσιάσουμε και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν ως προς τις ανακοινώσεις για σήμερα και ε, τώρα θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το εργαστήριο το οποίο διοργανώνεται από το θεματικό τμήμα Β με θέμα τις μακροπεριφερειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι επενδύουμε αρκετό χρόνο για τις εκθέσεις που αφορούν τις μακροπεριφερειακές ε, στρατηγικές και ε, Έχουμε και μία έκθεση εφαρμογής, η οποία είναι εξελίξη. Ο κύριος Κοτσολίνο είναι ο αρμόδιος εισηγητής και γι' αυτό και ε, διοργανώθηκε και αυτό το εργαστήρι, το οποίο θα ε, μας δώσει και κάποιες περισσότερες πληροφορίες ε, για τις ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές στην Ευρώπη. Να περάσω λοιπόν απευθεία στο πρόγραμμα για να μην ε, σας καθυστερώ και θα ήθελα να καλωσορίσω τους ομιλητές. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, είναι χαρά μας ε, να σας έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του εργαστηρίου. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, έννοιες, εξέλιξη και προκλήσεις καθηγητή Στέφαν Γκέσλε, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας, από την Νορβηγία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα σηκωθώ και λίγο για να με δείτε. Εγώ είμαι εδώ που με βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, δώσατε σε μένα την δυνατότητα και στους υπόλοιπους του πάνελ να ε, λάβουν σήμερα το λόγο. Ε, θα μου δοθεί φαντάζομαι η δυνατότητα να παρουσιάσω και κάποιες δικές μου επιστημονικές απόψεις επί του θέματος. Ελπίζω να μην είναι όλα αυτά ε, βαρετά. Σκέφτηκα να παρουσιάσω λιγάκι το τι ακριβώς συμβαίνει με το σχεδιασμό, με τις εξελίξεις ε, και ορισμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το μακροοικονομικό μακροπεριφερειακό εγχείρημα. Αυτή είναι η ε, ομιλία μου. Ε, ασχολείται βέβαια με κάποια ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχω διεξαγάγει με συναδέλφους και τα οποία εντάσσονται σε ένα βιβλίο το οποίο πωλείται και εμπορικά στο εμπόριο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ας δούμε λιγάκι στο παρελθόν να διερωτηθούμε γιατί να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Γιατί να εξετάσουμε τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και νομίζω ότι υπάρχουν ε, καταρχήν δύο ε, βασικοί και ενδιαφέροντες λόγοι. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές κατά κάποιον τρόπο εξετάζουν το θέμα της βέλτιστης ε, ρυθμιστικής περιφέρειας όπως το αναφέρουν και οι Ιταλοί, ο κύριος Μαγιώνε πιο συγκεκριμένα, ε, που ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ μεγάλη για να κρίνεται ως η βέλτιστη ρυθμιστική περιφέρεια στη Μεσόγειο, στη Βαλτική. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίε να είναι πιο στοχευμένε, πιο συγκεκριμένες. Μία άλλη βασική έννοια την οποία παρουσιάζει ο κύριος Κλάους Λέγκεβι, Γερμανός, είναι ότι οι προσπάθειες όπως το να υπάρξουν μακροπεριφερειακές ενώσεις, παραδείγματο χάρη είναι η Ένωση της Βαλτικής Θάλασσας, ο ίδιος το προτείνει αυτό, αυτές μπορούν να είναι ο κρίκος που θα προκαλεί την επαφή με τους πολίτες και παράλληλα θα γίνεται λόγος και για την ανάγκη ε, διεθνούς συνεργασίας, αλλά σε ένα μικρότερο πλαίσιο. Ας δούμε τώρα λιγάκι ε, τι σημαίνει μακροπεριφέρειες. Ε, βεβαίως, ως έννοια υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις, παρόλα αυτά όμως, αν δει κανείς την ε, γεωγραφία, την οικονομία, την πολιτική. Χρησιμοποιείται εμπρέως αυτή η έννοια με τρεις τρόπους. Καταρχήν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μία μακροπεριφέρεια. Ε, αυτό βέβαια σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η περιφέρεια Αζιάν είναι μακροπεριφέρειες σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά μπορούμε να το δούμε και κάτω από το πρίσμα της χώρας και να εντοπίσουμε μακροπεριφέρειες οι οποίες κατά κάποιον τρόπο είναι σε ενδιάμεση κλίμακα. Είναι ε, και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Και υπάρχει και ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 και παραθέτω είναι μια περιοχή, μια περιφέρεια η οποία ε, περιλαμβάνει διάφορες χώρες ή περιοχές ε, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσει που μπορεί να είναι στον τομέα των μεταφορών, του περιβάλλοντο και καθεξής. Σήμερα λοιπόν αυτέ όλε οι ανησυχίε έχουν προκαλέσει και μακροπεριφερειακές στρατηγικέ, δηλαδή ολοκληρωμένα πλαίσια τα οποία περιλαμβάνουν χώρε ε, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ε, που αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσει πολύ συχνά περιβαλλοντική φύσεω. Αυτό συμβαίνει, χάρη, στη Βαλτική θάλασσα, στο Δούναβι και αλλού. Και αυτό θα το δούμε και συνεχεία. Όλες αυτές βασίζονται σε πέντε βασικές αρχές, δηλαδή στην ενσωμάτωση, στο συντονισμό, στην συμπερίληψη των πολιτικών, στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει ως στόχο να επιτυγχάνει καλύτερο συντονισμό ε, σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αν προσπαθεί κανείς να συντονίσει όχι μόνο σε ένα επίπεδο, όχι μόνο οριζόντια δηλαδή, αλλά και κάθετα. Να υπάρχει κάθετο συντονισμό σε διάφορες χώρες. Αυτό πραγματικά είναι δύσκολο, είναι πρόκληση. Σήμερα, ε, κατά κάποιον τρόπο, εξακολουθούμε να έχουμε τα τρία όχι που βασικά ε, ήταν ε, μια συμφωνία ε, που χαρτίζεται όμως από όχι επιπρόσθετη χρηματοδότηση, όχι επιπρόσθετη θεσμή, όχι επιπρόσθετη νομοθετική διαδικασία. Πάντως προέκυψαν κάποιες ενώσεις και κάποια μορφή διαχείρισης στην μακροπεριφέρεια. Αυτό κατά κάποιον τρόπο διαχωρίζεται από άλλες προσπάθειες και άλλα εγχειρήματα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι όλα αυτά δημιουργούν σύγχυση, ότι είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν μία σειρά θεμάτων. Αλλά εν πάση εντοπίστηκε ότι υπάρχουν προεκτάσεις. Και πολύ συχνά αυτό ε, λόγω των... Ε, ε, επιπτώσεων και προεκτάσεων που προέκυψαν από τις, από τις συζητήσεις. Αυτό δηλαδή που μας καλέσετε και εσείς ε, σήμερα να κάνουμε είναι να δούμε κατά πόσον αυτές οι στρατηγικές μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να απαντήσω και σε αυτήν την ερώτηση, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε λιγάκι ιστορικά το τι συνέβη και να δούμε ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές δεν αφορούν μόνο την περιφερειακή συνεργασία με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς και έχουν άμεση σχέση με τη συνοχή, αλλά αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι ότι εδώ γίνεται περισσότερο λόγος για παραδοσιακές μορφές της περιφερειακής ε, ένταξης και ολοκλήρωσης είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εγώ βέβαια έρχομαι από την Νορβηγία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την Νορβηγική την Βόρεια Ένωση εμείς έχουμε και τη συνεργασία της Βαλτικής θάλασσας. Είναι μια ε, μακρά ε, συνεργασία, χρονικά μακρά, που ξεκίνησε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σταμάτησε βέβαια μετά τη συγκρούση Ανατολής ε, Δύσης. Και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθεί να διαμορφώσει αυτή την περιφερειακή συνεργασία στην επικράτειά της. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπίζουμε την μακροπεριφερειακή στρατηγική στρατηγική ως ένα εργαλείο ε, να χαρακτηρίσουμε την περιφερειακή συνεργασία και να εξετάσουμε και διάφορα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να σας ε, παρουσιάσω. Βλέπετε εδώ κατά κάποιον τρόπο ένα χάρτη της περιοχής. Ε, να πω το εξής, ότι την, τις μακροπεριφερειακές ε, συνεργασίες θα πρέπει να τις έχουμε ως ένα είδος ε, governance μιας διακυβέρνησης, αλλά και ως ένα είδος πειραματικού τρόπου για να δοκιμάσουμε νέες πολιτικές και νέες προσεγγίσεις. Είναι λίγο δύσκολο να τα δείτε αυτά στη διαφάνεια, αλλά παρόλα αυτά ε, βλέπετε ότι στην διαφάνεια βλέπουμε έναν κύκλο την πειραματική διακυβέρνηση μια προσπάθεια ε, να χαρακτηριστεί ας πούμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο όπου σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να έχουν ένα κοινό ευρύτερο πλαίσιο ε, στον τομέα της πολιτικής ε, παρά να εκχωρούν αρμοδιότητες σε τοπικές μονάδες, μονάδες δηλαδή κράτη-μέλη ή περιφέρειες που ε, μετά και αυτά, αυτές οι μονάδες ε, θα είναι αναγκασμένες όμως να λογοδοτήσουν και να βελτίσουν, βελτιώσουν το σύστημα της ε, διακυβέρνησης. Άρα το πειραματικό κατά κάποιο τρόπο δεν είναι πια πειραματικό γιατί έχει δοκιμαστεί. Αυτό είναι βασικά και το μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω ότι τουλάχιστον από ακαδημαϊκή σκοπιά θα πρέπει να επιτρέψουμε να εξεταστούν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και να δεχτούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον είναι πειραματικές αυτές οι προσπάθειες. Που σημαίνει βασικά ότι ως ένα κοινό πλαίσιο το οποίο έχει συμφωνηθεί και ακόμα και έχει προκληθεί από τα κράτη-μέλη πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Στρατηγικές ε, κρατών μελών ε, που ε, παίζουν σημαντικό ρόλο και ε, συμφωνούν ε, τα κράτη-μέλη για την πολιτική που πρέπει να χαράξουν και μετά ε, εκχωρούν αρμοδιότητες σε εθνικές μονάδες. Έχουμε λοιπόν συντονιστές που ασχολούνται με συγκεκριμένες προτεραιότητες και αυτοί έχουν ε, και κάποια ελευθερία για το πώς θα εφαρμόσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένες τομείς και μετά αναφέρονται. Αυτή λοιπόν είναι η γενική ιδέα. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ότι όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα ε, και ίσως είναι περίπλοκα, αλλά παρόλα αυτά να δείτε ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα για το πώς μπορεί κανείς να δοκιμάσει νέες μορφές της ε, υπερεθνικής ε, συνεργασίας, ε, συνεργασία ορισμένων κρατών μελών με συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία διαφέρουν από άλλες περιφέρειες. Ας πάρουμε ας πούμε τη Βαλτική και ας τη συγκρίνουμε με την Αδριατική ή την περιφέρεια του Ιωνίου. Έχουμε προτεραιότητες και αυτή η εικόνα δείχνει και άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο της συνεργασίας στο πλαίσιο της μακροοικονομικής στρατηγικής. Δεν πρόκειται μόνο για συγκεκριμένες στρατηγικές. Σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το συγκεκριμένο πείραμα είναι ότι μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκριση. Άρα δηλαδή μπορεί κανείς πολύ εύκολα να κάνει τη σύγκριση ανάμεσα σε διάφορες μακροοικονομικές στρατηγικές, το τι γίνεται, το πώς γίνεται και μπορεί να υπάρξει και ε, αμοιβαία συνεργασία και να μάθει κανείς πράγματα από τις διάφορες ε, αυτές ε, στρατηγικές. Τα κράτη-μέλη μπορούν δηλαδή να ζητήσουν και άλλα παραδείγματα. Ας πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα που θέλω να προβάλλω. Είναι οι προκλήσεις, οι δυσκολίες. Ε, να δούμε πώς είναι δυνατόν να ε, έχουμε μια καλύτερη εικόνα των προεκτάσεων. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να υπάρχει εξολόγηση αντικτύπου σε αυτές τις ε, στρατηγικές και θα ήθελα να παραθέσω την ειδική έκδοση του ε, Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αντιμετώπιση του ευτροφισμού στη Βαλτική θάλασσα. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν προεκτάσεις ε, ίσως όμως να χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο για να σας τα παρουσιάσω αυτά. Και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συνεργασίας ε, ανάμεσα στους ε, θεσμούς. Πλέον δεν μιλάμε για πειραματισμούς, μιλάμε για πιο μόνιμη συνεργασία, όπως ενώ χάρη το Φόρουμ Αλίας της Βαλτικής Θάλασσας. Όπως όλοι σας γνωρίζετε, οι μακροοικονομικές στρατηγικές έχουν ενταχθεί ως ε, ένα στοιχείο σε πολλές πολιτικές. Αυτά όμως ακόμα δυστυχώς παραμένουν στα χαρτιά και το θέμα είναι ε, πώς μπορούμε να τα εντάξουμε καλύτερα στα διάφορα ταμεία που υπάρχουν. Βεβαίως παραμένει η δυσκολία ε, της συνεργασίας, το σύστημα είναι περίπλοκο, αλλά για συγκεκριμένους φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόσο μάλλον για τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό είναι το θέμα που πρέπει να εξετάσουμε και να επιλύσουμε. Υπάρχει και κάτι άλλο. Οι εταίροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσονται με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν κάποιες στρατηγικές, από αυτό βέβαια δεν δημιουργεί πρόβλημα στη Βαλτική θάλασσα, παραδείγματος χάρη. Η Νορβηγία κατά κάποιον τρόπο ε, εντάσσεται Υπάρχουν διαφορές με άλλες στρατηγικές, παραδείγματος χάρη περίπτωση του Δουνάβεως, όπου έχουμε διάφορες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, προσβλέπουν στο να ενταχθούν, όπως είναι η Σερβία, αλλά και περιφέρειες ε, που δεν θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Ουκρανία. Ε, παρόλα αυτά όμως μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη στρατηγική. Και μετά υπάρχει και το θέμα των διακυβερνητικών φορέων όπως το Συμβούλιο των κρατών της Βαλτικής θάλασσας που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και μπορεί κανείς και να ισχυριστεί ότι αυτή η κλασική μορφή περιφερειακής συνεργασίας αυτή γίνεται όλο και περισσότερο υποστηρικτή Τη στρατηγική και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι σαφέ ότι η επιτυχία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε τελική ανάλυση εξαρτώνται και από την πολιτική βούληση των χωρών που συμμετέχουν. τελειώνοντα. ελπίζω να ήμουν σαφής στο ότι πρέπει κανεί τι μακροπεριφερειακές στρατηγικέ, να τι αντιμετωπίζει ω πειραματικέ με κανονικέ ε, προεκτάσει και αντικτύπου, ε, σε ορισμένε περιπτώσει, κάποιε στρατηγικέ να είναι πιο όριμε και όμως πράγματι είναι απαραίτητο να γίνουν μετρήσεις, να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει βελτίωση ε, με βάση συγκεκριμένους στόχους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οι μακροοικονομικές στρατηγικές αυτό που έχουν στόχο είναι να ξεκινάει η συνεργασία σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας ε, σημαντικός στόχος από μόνος του. Οι μακροοικονομικές στρατηγικές διαφέρουν από τις ε, πολυεπίπεδες στρατηγικές ε, που δεν έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται για πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε, μικρότερο, σε μικρότερη κλίμακα βασίζονται στην ε, καλύτερη συνεργασία. Επίσης αναφερθήκα στο ότι η συνεργασία θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να συγκρίνουμε την μακροπεριφερειακή συνεργασία, κάτι που δεν είχαμε κατά το παρελθόν, όπου είχαμε μόνο ε, την συγκεκριμένη ε, συνεργασία σε επίπεδο κυβερνήσεων, αυτό που ήταν ε, υπήρχε παραδείγματος χάρη στην Βαλτική. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα και μιλάμε για ε, καλύτερη συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Με αυτά, με αυτές μου τις παρατηρήσεις θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου και να προτείνω ότι αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι να μην αντιμετωπίζουμε αυτές τις μορφές στρατηγικής ως ένα απλό πρόγραμμα ε, υπερεθνικής συνεργασίας, διασυνοριακής συνεργασίας. Δεν είναι αυτό, είναι κάτι παραπάνω. Πρέπει να δούμε το πώς είναι δυνατόν ε, να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία που έχει σχέση και με διάφορα υπουργεία. Και τέλος, πρέπει να έχουμε κατά νου τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Και τέλος πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι βουλευτές μπορούν και αυτοί να αναλάβουν συγκεκριμένες λειτουργίες στο να ελέγχουν αυτό που ελπίζουμε ότι θα είναι η επιτυχία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και σχόλια, αλλά θα συνεχίσουμε με τις παρουσιάσει και θα κρατήσουμε τις ερωτήσεις για το τέλος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιαρμουλκάιτε. Ελπίζω να το πρόφερα σωστά. από το Τμήμα Πολιτικής Συνοχής του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και θα μας ε, μιλήσει για την συμμετοχή των διαρθρωτικών και επενδυτικών ε, ταμείων ε, στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα να σας παρουσιάσω την εμπειρία της Λιθουανίας κατά την εφαρμογή της στρατηγικής για την Βαλτική θάλασσα. Εγώ εργάζομαι για το Υπουργείο Οικονομικών της Λιθουανίας που είναι υπεύθυνο, το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση των διαδοτικών ταμείων. Εγώ ε, είμαι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό. Κατά την περίοδο 14 έως 20 μία από τις ευθύνε μου ήταν ε, να προσπαθήσω να συνδέσω με το εθνικό σύστημα ε, την στρατηγική ε, την, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βαλτική θάλασσα. Έχω χωρίσει την παρουσίασή μου σε δύο τμήματα. Καταρχάς θα ε, σας πω τι κάναμε για να ενσωματώσουμε στο σύστημά μας τη στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα. Θα σας δείξω κάποια αποτελέσματα της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και μετά θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποιες σκέψεις ως προς τον εντοπισμό των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και για τις ε, συστάσεις ε, για βελτιώσεις. Θα ήθελα για λόγους να σας παρουσιάσω καταρχάς κάποια εθνικά στρατηγικά έγγραφα ε, των ε, διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Στη Λιθουανία έχουμε μια συμφωνία σύμπραξης που καλύπτει πέντε τέτοια ταμεία και τρία επιχειρησιακά προγράμματα. Ένα για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου, ένα για την αλληλεία και για το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγώ θα ήθελα να σας αναφερθώ καταρχάς στο θέμα που αφορά τη συνοχή. Κατά την προετοιμασία της περίοδου 2014-2020. κάναμε μεγάλες προσπάθειες να συμπεριλάβουμε τη στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα στα εθνικά ε, έγγραφα, στρατηγικά μας έγγραφα. Έχουμε πολλές, πολλούς, ε, πολλές, πολλούς διακανονισμούς που αφορούν για παράδειγμα την αξιολόγηση και άλλα ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη Βαλτική ε, θα σας πω ότι θεωρούμε ότι πρέπει να έχει ως χαρακτηριστικό ένα πρόγραμμα για να συμμετέχει σε αυτή τη στρατηγική, για να συμβάλλει. Πρώτον, πρέπει να, έχει, να είναι σχετικό με τους τομείς πολιτικής, τις οριζόντιες, αρχές, δράσεις ή να είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα και επίσης πρέπει να υπάρχουν διεθνείς εταίροι. Να τις θυμάστε αυτές τις δύο προϋποθέσεις γιατί είναι σημαντικές και θα είναι πιο σημαντικές όταν θα μιλήσουμε για τα θέματα παρακολούθησης. Στην ε, Λιθουανία ε, βλέπουμε ότι υπάρχει σχέση και με το θέμα των, του περιβάλλοντος, της, ε, των μεταφορών και της ενέργειας και την αύξηση της ευημερία με τις επενδύσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην αποσχόληση. Στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα έχουμε εντοπίσει τους, ε, τις θεματικ, θεματικούς τομείς ε, που πρέπει να είναι τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού μας προγράμματος. Ε, οι επενδύσεις λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν κυρίως την ενέργεια, την καινοτομία και τις μεταφορές και λιγότερο τους κινδύνους, την ασφάλεια και την εκπαίδευση. Αυτός ο εντοπισμός των βασικών τομέων μας επιτρέπουν να δούμε μια ευρύτερη εικόνα των πιθανών ε, τομέων συνεργασίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια άλλα projects δεν μπορούν να συμβάλλουν σε άλλους ε, τομείς, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ή η υγεία. Στην εθνική μας νομοθεσία ε, έχουμε κάποιες διατάξεις που είναι φιλικές προς τη στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ε, επιπλέον ε, χρηματοδότηση, να χρησιμοποιήσουμε κάποιες οικονομίες για την συνεργασία με διεθνείς εταίρους στα πλαίσια προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας. Επίσης μπορούμε ένα τμήμα της χρηματοδότησης να δαπανηθεί εκτός του πλαισίου του επιχειρησιακού προγράμματος. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι διατάξεις ε, δίνουν μια πολύ καλή βάση για, τις ε, διασυνοριακές, ε, για τα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα εφαρμογής, έχουμε κάποια κριτήρια επιλογής που δίνουν ε, προτεραιότητα στα projects τα οποία ε, συμβάλλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής. Πέντε μέτρα ήταν ο γνωμονά μας, ε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό μέτρων, δείχνει παρόλα αυτά μια σημαντικότερη εστίαση στη στρατηγική. Επίσης, έχουμε κάποιες απαιτήσει των θεσμικών μας οργάνων να εντοπίζεται κατά πόσο τα προγράμματα και με ποια μέτρα συμμετέχουν στη στρατηγική. Έχουμε και οι ίδιες προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για τους ενδεχόμενους υπευθύνου έργων, των project managers, ε, για τα προγράμματα που θέλουν να εφαρμόσουν, τι προστιθέμενη αξία έχουν σε σχέση με την στρατηγική για τη Βαλτική. Αυτό μας βοηθά στο να αυξήσουμε ε, την ε, ευαισθητοποίηση τη θεσμική αλλά και των υπευθύνων έργων ε, ε, δεν είναι πάντοτε εντελώς ακριβής η αξιολόγηση. Τα μέτρα μερικές φορές είναι πολύ περίπλοκα και όλα τα, μέτρα, ε, υπό όλα τα προγράμματα υπό το συγκεκριμένο μέτρο δεν συμμετέχουν υποχρεωτικά ε, στη στρατηγική. Επίσης, μερικές φορές δεν υπάρχουν και οι απαραίτητες ικανότητες από πλευράς υπευθύνων έργων για τη συμβολή στην στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα παρακολούθησης των των Δεν έχουμε βέβαια ξεχωριστό ε, σύστημα για τη συγκεκριμένη στρατηγική για τη Βαλτική. Έχουμε λοιπόν ε, συμπεριλάβει ε, μια ειδική καρτέλα στο πλαίσιο της στρατηγικής που μας επιτρέπει να κάνουμε έναν υπολογισμό της συμβολής των προγραμμάτων σε αυτήν, σε ε, δύο ε, επίπεδα. Πρώτα, ε, κάνουμε μία μέτρηση της θεματικής συμβολής, αν είναι σχετική δηλαδή, αν καλύπτει οριζόντια θέματα. Επίσης, κάνουμε έναν υπολογισμό της διασυνοριακής διάστασης και επίσης του κατά πόσο υπάρχει συνεργασία με έναν διεθνή εταίρο. Αυτό βέβαια έχει διευκολύνει πολύ τη διαδικασία παρακολούθησης, ειδικότερα σε σχέση με το τι συνέβαινε το 2017 έως 2013, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δείξουμε έναν εντυπωσιακό αριθμό διασυνοριακών προγραμμάτων, αλλά αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να εντοπίσουμε ενδεχόμενους τομείς διασυνοριακής συνεργασίας. Δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτή τη διαφάνεια που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες προώθησης συνεργασίας πάντως και η Λιθουανία ε, συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό ε, στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, και ήταν επίσης συντονίστρια στην βιοοικονομία υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συμμετέχουμε επίσης ενεργά στις θεματικές δράσεις για το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θέλουμε να ισχύουμε τη συμμετοχή σε ε, διεθνή συνεργασία. Στα, στη διαφάνεια αυτή μπορείτε να δείτε κάποια αριθμητικά στοιχεία για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Από την αρχή αυτής, για όλα τα προγράμματα που ξεκίνησαν την εφαρμογή τους, περίπου 27% θεωρείται ότι συμμετέχουν στη στρατηγική ε, για την ε, περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Αυτό το ποσοστό όμως δείχνει απλώς ε, μία θεματική συμβολή. Τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την συνοριακή συνεργασία παρουσιάζουν μείωση. Έχουμε δαπανίσει 2,3% των τριών ε, ε, διαρθρωτικών και επενθετικών ε, ταμείων. Τα προγράμματα αυτά αφορούν κυρίως την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, την ενέργεια και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν βλέπουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά, προφανώς το ερώτημα είναι για ποιο λόγο ο όγκος ε, των προγραμμάτων για τη συνεργασία δεν έχει αυξηθεί εφόσον υπάρχουν όλες οι νομικές διατάξεις και το ε, απαραίτητο περιβάλλον. Προφανώς υπάρχουν κάποια σημεία συμφόρησης. Θα ήθελα σήμερα να αναφερθώ σε τρία από αυτά. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να βρούμε πολύ περισσότερες προκλήσεις. Ο καθένα από εμά θα μπορούσε να έχει μια ιδέα για μια ενδεχόμενη πρόκληση, αλλά ας επικεντρωθούμε σε αυτά. Καταρχάς, πολύ λίγοι γνωρίζουν τη στρατηγική για τη Βαλτική ε, θάλασσα. Μόνο 14% σύμφωνα με μελέτη του Ευρωβαρομέτρου ε, με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου γνωρίζουν ε, την στρατηγική αυτή και σε σχέση με άλλες μακροπεριφερειακές στρατηγικές αυτό το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο. Επίσης δεν υπάρχει θεσμική ευαισθητοποίηση. Δηλαδή οι θεσμοί μας δεν γνωρίζουν, ε, πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν την στρατηγική για την Βαλτική Θάλασσα, δεν βλέπουν τα ωφέλη της και δεν πιστεύουν στην προστιθέμενη αξία της. Πώς λοιπόν κάποιος που έχει την δύναμη να επιφέρει την αλλαγή, πώς θα το κάνει, πώς θα είναι αποτελεσματικός επιφέροντας την και αυτή αν δεν πιστεύει στη στρατηγική. Επίσης, η πρόσφατη εμπειρία μου όσον αφορά την ε, διαχείριση των, ε, του δικτύου των αρμοδίων αρχών για τη στρατηγική έδειξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η διάφο, διαφορετική εφαρμογή μεταξύ των χωρών που είναι πολύ δύσκολο να ε, συνδυαστεί. Θα ήθελα να κάνω και τρεις συστάσεις βάσει αυτών που σας παρουσίασα για τα σημεία συμφόρησης. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, πρέπει να αυξήσουμε την ορατότητα της ενωσιακής στρατηγικής για τη Βαλτική θάλασσα. Να σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα της πολιτικής συνοχής στη Λιθουανία. Στη Λιθουανία η πολιτική αυτή είναι πάρα πολύ επιτυχής, ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους πολίτες μας πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι πάνω από 90% των ε, Λιθουανών ε, γνωρίζουν ε, την πολιτική συνοχής και 6 από τους 10 ερωτηθέντες είπαν ότι έχουν προσωπική εμπειρία του ωφέλου αυτών των επενδύσεων 14% μιλούν υπέρ της ε, στρατηγικής και 90% υπέρ της πολιτικής συνοχής, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι πρέπει να αυξήσουμε την ορατότητα και των εργαλείων της διασυνοριακής μας συνεργασίας. Έχουμε πλατφόρμες, έχουμε ιστοτόπους ε, για την αναζήτηση εταίρων, όμως πολύ λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τη διαδικασία. Ε, ε, μία δεύτερη σύστασή μου είναι να είναι αναπόφευκτη αυτή η στρατηγική για τη Βαλτική θάλασσα. Σας ανέφερα τις προϋποθέσεις ε, που έχουμε θέσει για τους θεσμούς μας και τους υπευθύνου έργων να αναγνωρίσουν κατά πόσο συμβάλλουν τα προγράμματά τους, τα έργα τους στη στρατηγική αυτή. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και των θεσμών. Βέβαια η ευαισθητοποίηση δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, ε, γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση, αλλά πιστεύω ότι το να προχωρά κανείς αργά είναι καλύτερα από το να μην προχωρά καθόλου. Και κάθε φορά που με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτούν κάτι για τη στρατηγική αυτή, το θεωρώ μία μικρή νίκη προς ε, έναν ε, ευρύτερο στόχο. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τη διασυνοριακή συνεργασία. Σας έδωσα μόνο ένα παράδειγμα προηγουμένω. Μπορώ να πω πολλά άλλα παραδείγματα ε, για επιπρόσθετη χρηματοδότηση μέχρι ε, ωφέλη που δεν αφορούν τη χρηματοδότηση. Όμως οι ενδεχόμενοι υπεύθυνοι έργων πρέπει να πιστεύουν ότι υπάρχει όφελο στο μέλλον από τι προσπάθειε που κάνουν σήμερα. Επίσης, μία ακόμη για την ευελιξία και την απλοποίηση των κανόνων. Πολύ το αναφέρουμε αυτό κατά την ε, προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περίοδου και πιστεύω ότι η διασυνοριακή συνεργασία είναι ο τομέας στον οποίο χρειαζόμαστε απλούς, σαφείς και ευέλικτου κανόνες που είναι εύκολο να συνδυαστούν, που προάγουν την συνεργασία χωρί να την παρακολύουν, χωρί να την επιβαρύνουν, Οπότε το λέω αυτό σε σχέση με την προετοιμασία ε, των προτάσεων από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και προ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όσον αφορά τι διαπραγματεύσει. Και για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να σα πω ότι ο κόσμος της στρατηγικής για τη Βαλτική θάλασσα πέχει πολύ από την τελειότητα. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις αλλά και ε, πολύ μεγάλο δυναμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί με κοινέ προσπάθειες. Θα ήθελα λοιπόν να ε, σας ευχηθώ να είμαστε όλοι φιλόδοξοι, να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε, να επιφέρουμε την αλλαγή που θέλουμε. Βλέπετε εδώ ε, τα στοιχεία μου για να έρθετε σε επαφή μαζί μου αν θέλετε να υποβάλλετε περισσότερες ερωτήσεις ή να λάβετε περισσότερη πληροφόρηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Φέλιξ Μολτοβάν ο οποίος ε, θα μας παρουσιάσει την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, ε, προοπτικές μετά το 2020. Ο κύριος Μολτοβάν θα μιλήσει εξ ονόματος της Ουγγρικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εμπειρία μα από την εφαρμογή της στρατηγικής ε, του Δούναβη. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτά τα οποία θα πω δεν αποτελούν ε, το σύνολο τη συνένεση για τη στρατηγική, αποτελούν την εμπειρία της ουγγρική εφαρμογή. Τώρα, είναι πολύ δύσκολο ε, να μιλά κανείς για το μέλλον, ε, ακόμα και όταν τα πράγματα βαίνουν ομαλώς. Αλλά οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κάνουν τα πράγματα όλο ένα ε, και πιο δύσκολα και τις προκλήσεις μεγαλύτερες. Έχω απαριθμίσει εγώ κάποια στοιχεία, κάποιες πτυχές που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες προκλήσεις. Έχουμε το Brexit καταρχάς, το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει την πολιτική συνοχή μετά το 2020 τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εξέδωσε και πέντε έγγραφα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν ε, πολλές και ποικίλε δυνατότητες που θα μπορούσαν να επιλέξουν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, με τόσες πολλές μεταβλητές, οι οποίες καθορίζουν ε, την μακροπεριφερειακή στρατηγική και ε, για πιο λίγο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ε, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Βέβαια θα μπορούσα να πω ότι η πιο παλιά μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι μόνο 8 ετών, που σημαίνει ότι το να έχουμε μία ε, στρατηγική που περιλαμβάνει τόσους πολλούς εταίρους και τόσους πολλούς παράγοντες που να λειτουργεί αποτελεσματικά δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα. Ε, επειδή όμως το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πρώτον πυλών, πιστεύω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα και να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Ε, ξεκίνησα την παρουσίασή μου δίνοντάς σας ε, κάποια στοιχεία για το πώς ε, βλέπουμε εμείς ε, την παρούσα εφαρμογή της στρατηγικής της περιοχής του Δούναβη. Όλοι γνωρίζουν τα τρία όχι, τα οποία καθοδηγούν την εφαρμογή. Δεν υπάρχουν ε, νέα νομοθεσία, δεν υπάρχει εμπλοκή των, για πολιτικά κίνητρα και δεν υπάρχουν και νέα κονδύλια. Ε, καταλαβαίνω το σκεπτικό, αλλά κατά την άποψή μας αυτά τα τρία όχι οδήγησαν τελικά σε τρία διαφορετικά όχι, τρεις διαφορετικές αρνήσεις που σημαίνουν δεν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα, δεν υπάρχει προβολή και δεν υπάρχει και αίσθηση της ιδιοκτησίας ε, ε, αυτών. Μπορεί να φαίνεται πολύ αυστηρό αυτό, αλλά σε επίπεδο εφαρμογή, δυστυχώ αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι η πολιτική όθηση ε, έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται και αρκεί κανείς να δει τι συμμετοχή έχουμε ε, σε επίπεδο υψηλών πολιτικών προσώπων στις αιτήσιες ε, συνεδριάτηση και βλέπουμε ότι τα πράγματα φθήνουν. Όσον αφορά την προβολή, ε, διαπιστώσαμε ότι πολλά επιχειρησιακά προγράμματα εντό τη Ουγγαρίας δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει μακροπεριφερειακή στρατηγική. Ε, κάτι το οποίο είναι ατυχέ, διότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική θα μπορούσε να του ε, προσφέρει ένα στρατηγικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να δαπανώνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να τους υποδείξει και να να τα δαπανούν πιο αποτελεσματικά. Όσον αφορά τώρα την ιδιοκτησία, αυτό το οποίο ισχύει και για τη συμμετοχή είναι ότι βλέπουμε ότι και σε επίπεδο διευθύνουσας επιτροπής ε, για το Δούναβι δεν έχουμε ίση εκπροσώπηση από όλες τις χώρες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες κάνουν μια προσπάθεια ε, και είναι παρούσες σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις επιτροπής, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη μείωση στη συμμετοχή. Και αυτό σίγουρα αποτελεί πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε εάν θέλουμε οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές να ε, ε, χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Τώρα, επειδή υπάρχουν όλα τα παραπάνω και κυρίως επειδή δεν υπάρχει πολιτική στήριξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, εξακολουθούν να είναι μέσα τα οποία είναι πάρα πολύ ήπια. Από τη μια αυτό το αντιλαμβάνομαι, διότι στην περίπτωση της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη, η δομή της στρατηγικής είναι πάρα πολύ σύνθετη. Υπάρχουν εθνικοί συντονιστές, υπάρχουν μέλη της Διευθύνουσας ε, Επιτροπής, υπάρχουν συντονιστές ε, των προτεραιοτήτων της Διευθύνουσας Επιτροπής και το να πλασάρουμε αυτή την ιδέα της μακροπεριφερειακής στρατηγικής και να πείσουμε κάποιον ο οποίος δεν συμμετέχει ότι όντως υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στη συμμετοχή, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ιδιαίτερα δύσκολο. Μια άλλη πρόκληση της περιοχής του Δούναβη είναι ότι περιλαμβάνει κάποιες προτεραιότητες οι οποίες αποκλείουν πολύ μεταξύ τους. Ε, υπάρχει για παράδειγμα η Βάδη Βιτεμβέργη από τη μια πλευρά της ε, ε κλίμακας και έχουμε και τη Μολδαβία από την άλλη πλευρά. Καταλαβαίνετε βέβαια όλοι ότι οι κατεπίγουσες προτεραιότητες των δύο περιοχών ε, είναι πάρα πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Και αν το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως βάση, θα αντιληφθείτε ότι ε, το να καταλήξουμε σε συνένεση μεταξύ των συμμετοχών ανεξάρτητα ε, του τι πρόκειται, πρόκειται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολύ μικρή η σχέση μεταξύ μακροπεριφερειακών στρατηγικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων. Όπω είπα και προηγουμένω, κάποια επιχειρησιακά προγράμματα δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Αφενός το αντιλαμβάνομαι αυτό και εξηγείται και εύκολα, διότι όταν ε, ε, διαπραγματευόμασταν τη στρατηγική της περιοχής του Δούναβη, κάποια, ε, αν όχι τα περισσότερα από τα επιχειρησιακά προγράμματα, είχαν ήδη αποφασιστεί και υπήρχε ήδη πλαίσιο. Αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον είναι να επαναληφθεί αυτό στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα σχολιάσω και στη συνέχεια. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε, το οποίο παρακολεί πάρα πολύ την εφαρμογή της στρατηγικής, είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των μέσων χρηματοδότηση και ε, αυτών που τα εφαρμόζουν. δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία κατά το χειρισμό των θεμάτων αυτών και αυτό επιβραδύνει και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων και την πρόοδο και παρακολεί και όλους εκείνους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποιες ιδέες και δεν μπορούν να ε, παρουσιαστούν και να παρουσιάσουν και να προτείνουν κάποια προγράμματα. Τελευταίο σημείο, η περιορισμένη συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ατυχές, διότι από την πολύ περιορισμένη εμπειρία που έχω εγώ από τι μακροπεριφερειακές στρατηγικέ, μπορούμε να αντλήσουμε πολλά διδάγματα ο ένα από τον άλλον. Πολλέ καλέ πρακτικέ θα μπορούσαμε να τι χρησιμοποιήσουμε και να τι εκμεταλλευτούμε, διότι όλε αυτέ οι στρατηγικέ έχουν περάσει από αυτέ τι διαδικασίε ε, τι οποίε θα αντιμετωπίσουν οι νέε στρατηγικέ. Ε, και η μεγαλύτερη λοιπόν ε, συνεργασία μεταξύ των στρατηγικών αυτών στο μέλλον θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Βέβαια δεν είναι όλα ζωφερά. Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλέ δυνατότητε για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, και σας έχω ετοιμάσει και δύο διαφάνειες με συστάσεις τις οποίες θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη. Μία από τι μεγαλύτερε προκλήσεις ε, για την οποία δεν έχω κάποια συγκεκριμένη σύσταση είναι πώς μπορούμε να δώσουμε πολιτικά κίνητρα. Πρέπει ε, να πείσουμε ε, τους πολιτικούς ε, να υποστηρίξουν αυτές τις στρατηγικές και να υπάρξει μια νέα όθηση για αυτή τη στρατηγική, διότι έτσι και μόνον έτσι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές για να επιλύσουν τις παρούσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν μια πολύ καλή πλατφόρμα για πιο τίμια και πιο άμεση επικοινωνία. Αλλά δυστυχώς δεν έχω δει να χρησιμοποιούνται αυτές οι στρατηγικές για να προτείνουμε λύσεις για την κρίση, για τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Η Ουγγαρία οργανώζει ένα ετήσιο φόρουμ τον Οκτώβριο και προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε κάποια θέματα στο ημερήσια διάταξη τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στην επόμενη περίοδο. Παραδείγματο χάρη, ασφάλεια εφοδιασμού και ανάπτυξη υποδομών στην ενέργεια, διαφοροποίηση για την ασφάλεια εφοδιασμού. Αλλά δεν έχω ε, δει και την άποψη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, ποιε θεωρούν πιο επίγουσε κρίσει ε, και δεν έχω δει και άποψη για τη μεταναστευτική κρίση που είναι πιο σημαντική. Ε, δίνεται και μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε και τις απόψεις των κρατών μελών που συμμετέχουν και να προσφέρουν και κάποιες λύσεις ε, για τις κρίσεις αυτές. Προκειμένου όμως να συμβεί αυτό, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, και να αποτελέσουν εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων, πρέπει να ξαναδούμε το σχέδιο δράσης και πρέπει να εξορθολογιστεί. Όπως σας είπα και προηγουμένως, Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σύνθετο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο σωστά στοχευμένο, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση που ανέφερε και η συνάδελφος από τη Βαλτική προηγουμένως. Τώρα, χρηματοοικονομικό σκέλος τι μπορούμε να βελτιώσουμε εδώ. Όπω σα είπα προηγουμένω, εάν συμπεριληφθούν οι μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ στο επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, θα έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Χωρί ε, χρηματοοικονομική υποστήριξη, οι μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικέ. Μόλι μου είπαν ότι πρέπει να τελειώνω, επομένω θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο Συγκεκριμένως Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για αυτό το θέμα. Μία πολύ πρακτική προσέγγιση και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ουγγαρία είναι να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα για τις ε, διαχειριστικές αρχές ε, των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εργάζονται στην Ουγγαρία, να μπορούν να συγκεντρωθούν όλοι μαζί και να δούνε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τη στρατηγική και πώς μπορεί η στρατηγική της περιοχής του Δύναβη να εξορθολογήσει τις δαπάνες τους και να είναι πιο αποτελεσματικές. Όσον αφορά το συντονισμό, το πρόγραμμά μας έχουμε μια δομή που λέγεται το τρίο των προεδριών. Αλλά ε, θα πρέπει να διαδραματίσει πιο στρατηγικό ρόλο αυτό το τρίο των Προεδρεών για να δει πώς θα μπορούσε να προχωρήσει το θέμα των στρατηγικών. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά οι προεδρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν κάθε χρόνο στο στρατηγικό πλαίσιο, συγγνώμη. Και επομένως ε, ε, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να καθορίσουμε πολιτικές προκλήσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσει ένα τρίο προεδριών όπως γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, δραστηριότητες επικοινωνίες. Εδώ χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειαζόμαστε ανθρώπους με καλά προγράμματα, ε, με πρόγραμματα τα οποία θα επιλύνουν τοπικά θέματα. Θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να αντιλαμβάνονται πώς δουλεύουν οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές για να έρχονται και σε εμά με ιδέες ε, τις οποίες θα μπορούμε στη συνέχεια ε, να τους βοηθήσουμε να τις εφαρμόσουν. Επίσης, λέω ότι οι εθνικοί συντονιστές θα χρειαστούν προπολογισμό το γεγονός ότι οι διάφορες χώρες δεν θεωρούν κτήμα τους αυτά τις στρατηγικές και κυρίως χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επειδή δεν μπορούν να ταξιδεύουν και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ε, έχουν ε, και έλλειψη παρουσίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να βοηθήσουμε αυτούς τους εθνικούς συντονιστές που δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει κάποιο προπολογισμό για να μπορούν να τους καλύπτουν τα ταξιδιωτικά τους έξοδα για να μπορούν να είναι παρόντες όταν λαμβάνονται αποφάσεις. Ε, διοικητικές δυνατότητες. Και εδώ θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα γιατί πολλές χώρες ε, ε, ε, ε απλώς ε, δίνουν σε κάποιο διπλωμάτι το επιπλέον καθήκον της συμμετοχή σε αυτή την επιτροπή. Για να υπάρχει όμως αποτελεσματικότητα θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες διοικητικές δυνατότητες και να βελτιωθούν σίγουρα. Πόσο χρόνο έχω? Δύο-τρία λεπτά ακόμα, ωραία. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Τι πρέπει να αποφύγουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτήσει ένα πάρα πολύ καλό έγγραφο για το παρόν επίπεδο εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών. Εμεί συμφωνούμε με τι περισσότερε ε, ιδέε που έχουν παρουσιάσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να σας ε, ε, επισημάνω. Υπάρχουν κάποιοι ε, τομείς προτεραιότητας οι οποίοι είναι εκ Δεν θεωρούμε ότι είναι καλή λύση αυτή. Ε, δεν μπορούν έτσι να είναι δραστήριοι οι ε, φορείς ε, με τομείς προτεραιότητες οι οποίοι αλλάζουν. Ε, αυτά κατά την άποψή μας δεν επιτρέπουν την καλή εφαρμογή. Επίσης, το να μην υπάρχουν κάποιοι τομείς προτεραιότητες και να τους διαγράψουμε τελείως, αυτό θα πρέπει να είναι η ίστατη λύση. Πριν φτάσουμε σε αυτό, θα πρέπει να έχουμε κάποιους τομείς προτεραιότητες, τους οποίους θα τους συμπεριλάβουμε πολύ καλύτερα στη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα και με αυτά θα ολοκληρώσω. Η εκπεριτροπή προεδρία είναι πολύ καλή ιδέα. Βλέπουμε ότι οι χώρες ε, περιμένουν τη στιγμή που θα αναλάβουν τα ενία και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει και το ετήσιο φόρουμ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ε, ε, σημαντικό γεγονός. Έχουμε ενδιαφερομένους κάθε χρόνο ε, που δείχνει ότι υπάρχει και ενδιαφέρον για τις αγροπεριφερειακές στρατηγικές. Επομένως τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε τι στοιχεία έχουμε, τι εμπειρία έχουμε και θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε λίγο ακόμα. Κάτι τελευταίο, η προσέγγιση μας όταν αναλάβουμε την Προεδρία ήταν να συμπεριλάβουμε και τις γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στρατηγική. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική του δύναμη μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ καλό ε, εργαλείο για την πολιτική διεύρυνση και γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινήσαμε μια σειρά από project στο παρελθόν, τα οποία ε, εγκρίθηκαν από το Διεθνές ε, ε, Πρόγραμμα του Δούναβη και έχω αναφέρει μόνο το κοινό πρόγραμμα ε, ΤΙΣΑ και το Σολοτβίνο πρόγραμμα, τα οποία περιλαμβάνουν και τις γειτονικές χώρες εκτός Ένωσης. Ε, και αυτό είναι ο μόνος τρόπος κατά την άποψή μας μπορούμε, ε, με τον οποίο μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτές τις χώρες ε, που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά συμμετέχουν στη στρατηγική για το δύναμο. μέσω κοινών προγραμμάτων για να μπορέσουν να βιώσουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι προσδοκίες υπάρχουν κλπ. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες και να τις εμπλέξουμε περισσότερο ε, να ενταχθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Αυτά λοιπόν. Ε, έχετε τις διαφανειές μου, ε, θα μπορούσα να συνεχίσω πραγματικά για πολύ περισσότερο. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ ελεύθερα, έχετε και τα στοιχεία ε, επικοινωνίας μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα και ελπίζω να σας δω όλους στις 18 και 19 Οκτωβρίου στη Βουδαπέστη για την έκτη ετήσια συνάντηση του Φόρουμ της ε, Περιφερειακής Στρατηγικής στο Δουναβή. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Φάβια, ο οποίος ε, είναι διευθυντής του, του Τμήματος Πολιτικών Συνοχής από την Ιταλία και θα μας παρουσιάσει μια άλλη μακροπεριφερειακή στρατηγική, τη στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο και την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την περιοχή των Άλπαιων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα σας μιλήσω εγώ για τις τελευταίες ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, και εγώ θέλω με την ομιλία μου να επικυρώσω όλα αυτά που υπάρχουν στο πρόγραμμα με στοιχεία. Έχουμε λοιπόν ε, μια άσκηση, διοικητική άσκηση σχετικά με την ε, αποτελεσματικότητα, αλλά εγώ θα ήθελα, όπως σας είπα, να επιβεβαιώσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου, γιατί ερχόμενος εδώ και ακούγοντας αυτά που είπαν, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία ε, και ορισμένα θέματα που ανέφεραν είναι πραγματικά ε, σημαντικά. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω πολλά από αυτά που ελέγχθησαν. Θα επιβεβαιώσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι μετά θα περάσω στα συμπεράσματά μου και θα αναφέρω τη δική μου άποψη. Γιατί κατά την άποψή μου ο διάβολος ε, κρύβεται στη λεπτομέρεια και βεβαίω επί στρατηγικής απόψεως σε αυτό το επίπεδο συμφωνώ με αυτά που λένε, αλλά ξέρετε στην πρακτική εγώ διαπίστωσα ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο χάλια και αν θέλει κανείς να τα αλλάξει πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικός γιατί οφείλει να αναλάβει και κάποιους ε, κινδύνους. Συμφωνώ απόλυτα όσον αφορά στην απλούστευση των κανόνων των κανόνων της χρηματοδότησης ε, του θεσμικού ρόλου. Οι μακροπεριφέρειες είναι μια καταπληκτική άσκηση για να ξεπεράσει κανείς κάποιες ακαμψίες του συστήματος. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε χώρες, σε κυβερνήσεις, φορείς. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι πρέπει η συνεργασία να επεκταθεί και στο πολιτικό και στο τεχνικό επίπεδο. Αυτά βέβαια να μην συγχέονται, γιατί εγκυμονούν κινδύνους. Το τέταρτο που είναι πιο σημαντικό είναι η προσαρμογή ε, και ο ευθυγραμμισμός των δραστηριοτήτων. Δεν αφαίρομαι μόνο στα γενικότερα προγράμματα, αλλά στα εθνικά, στα περιφερειακά και στα κονδύλια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για κάποιες μακροπεριφερειακές δραστηριότητες, μεταφορές, ε, ναυτιλία, όλο αυτό το σύστημα πρέπει να ευθυγραμμιστεί για να αποδώσει αποτελέσματα. Και αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα επί των οποίων συμφωνώ. Όσον αφορά τις ε, περιφέρειες, ε, θα σας ε, μιλήσω για την εμπειρία μου σε δύο περιφέρειες και θέλω να σας πω ότι η Ιόνια και το Ιόνιο με συγχωρείτε <laughs> και η Αντριατική περιλαμβάνουν τέσσερα ε, κράτη-μέλη και τέσσερα μη κράτη-μέλη. Είναι δύσκολες αυτές οι περιοχές, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μέχρι πριν από κάποια χρόνια στην περιοχή αυτή μενόταν ο πόλεμος. Είναι λοιπόν σημαντικός ο ρόλος που παίζουν όχι μόνο οι στρατηγικές, αλλά και οι πολιτικές πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν αμέσως μετά το πέρας του πολέμου με στόχο να επανέλθει ο διάλογος ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει το θέμα της οικειοποίησης αυτών των στρατηγικών. Ο διάλογος που υπήρχε κατά το παρελθόν είναι πολύ σημαντικός για να λυθούν προβλήματα της περιοχής. όλα αυτά όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν γιατί όπως βλέπετε στην περιοχή αυτή περιλαμβάνονται και το Κοσφοπέδιο και η Φύρομ. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά στην ε, μακροστρατηγική, έχουμε έναν ε, φορέα διαχείρισης ε, που εναλλάσσεται κάθε χρόνο και μάλιστα τώρα έχει οθετηθεί η τριμερής προεδρία έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επίση ε, υπάρχει και κοινή προεδρία. Αυτό για να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία με τις άλλες χώρες. Έχουμε θεματικές ομάδες οι οποίες κάνουν την τεχνική δουλειά και πρέπει να σας πω ότι αυτές οι ομάδες εστιάζονται ιδιαίτερα στο να εντοπίσουν τις ιδιαιτερότητες της ε, περιοχής και μετά ενδεχομένως να ε, εντοπίσουν ε, συγκεκριμένα προγράμματα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και άλλη και να γίνουν και άλλες αναλύσεις, διότι ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να λάβουν χώρα απλά και μόνο αναγνωρίζοντας ε, ποια είναι τα κοινά θέματα, τα κοινά προβλήματα σε αυτή την περιοχή. συνεδριωτική παραμύθος χάρη, υπεραλίευση. Και τι θα γίνει στην μεταγενέστερη περίοδο. Αν ας πούμε σταματήσει η Ιταλία την αλήψη θα κάνει η Κροατία. Τι γίνεται τώρα με την Γιουζέρ, με αυτή την περιοχή. Είναι ε, πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Ο διάλογος ε, έχει ξεκινήσει και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες ε, κατά το παρελθόν ε, είχαν εχθρικές σχέσεις τώρα πλέον έχουν κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Και βλέπω ορισμένε χώρες οι οποίες πριν από κάποια χρόνια, σας είπα, είχαν εχθρικές σχέσεις, τώρα συνεργάζονται. Γιατί έχουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν. Και η οικειοποίηση αυτής της ε, στρατηγικής ε, σίγουρα είναι, υπάρχει στις ε, χώρες μέλη, όχι τόσο σε αυτές που δεν είναι μέλη, αν και υπάρχει και κάποια κόπωση. διότι τα νέα κράτη-μέλη έχουν δυσκολία στο να συμμετέχουν, άρα δηλαδή στο θέμα της χρηματοδότησης κάτι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να φουσκώσει και το πορτοφόλι των νέων μελών και αυτών που δεν συμμετέχουν. Όπως σας είπα υπάρχει αυτή η Προεδρία με τρία κράτη και αυτό επιτρέπει ε, να υπάρχει καλύτερη συμμετοχή και τώρα μπορεί να υπάρχει και ηγετικός ρόλος και στις ε, τεχνικές ομάδες για να επιτευχθούν ε, αποτελέσματα. Οι τεχνικές ομάδες συνήθως ακολουθούν το δικό τους δρόμο και μιλάνε πάρα πολύ. Ε, δεν είναι δηλαδή στοχευμένες στο να επιτύχουν αποτελέσματα. Ως εκ τούτου ε, το Διοικητικό Συμβούλιο ε, έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνει και η αυτονομία των τεχνικών ομάδων. Και όπως σας είπα, θα πρέπει να γίνονται και συζητήσει σε θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα κονδύλια που υπάρχουν και οι κανόνες και οι δραστηριότητες ε, να είναι πιο αποτελεσματικές, να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και με τα εθνικά ταμεία, ε, ακόμα και τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άμεσα κονδύλια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί περαιτέρω διάλογος. Έτσι λοιπόν, κατά την άποψή μου, ο ρόλος της Επιτροπής ε, ε, και ο ρόλος της Επιτροπής είναι ο εξής. Είναι μια καλή προσέγγιση, αλλά ε, η Κομισιόν έχει αποσυρθεί από τη Συμπροεδρία ε, γιατί ακριβώ ε, την έχουν οικειοποιηθεί την Προεδρία τα κράτη-μέλη. Ο ρόλος της Κομισιόν όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός. Υπάρχει μία κόποση όσον αφορά τα κράτη-μέλη, κυρίως τα πρόσφατα κράτη-μέλη και τα μικρότερα κράτη-μέλη δεν κατανοούν ακριβώς τους, τις διαδικασίες και αυτό δεν είναι εύκολο να το μάθει κανείς ακόμα και για ε, πεπειραμένους ε, υπαλλήλους. Ο, ρόλος της Κομισιόν είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Τώρα, ας δούμε λιγάκι την ε, συνεργασία στην, περιοχή των Άλπων, Ιουζάλπ. Εδώ έχουμε κράτη-μέλη, οι τρεις από τις τέσσερις, είναι και ιδρυτικές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές που δεν συμμετέχουν, μάλλον που δεν είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ ισχυρέ χώρες. Και για αυτές δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο. Αυτό λοιπόν είναι ένα εγχείρημα ε, το οποίο είναι και η τελευταία μακροστρατηγική, μακροπεριφερειακή στρατηγική. Βέβαια, ορισμένε περιοχές θέλουν ε, να δείξουν ότι είναι αυτόνομες ε, και ως εκ τούτου θέλουν και οι περιοχές αυτές να έχουν την δυνατότητα να τεκμηριώσουν την άποψή τους. Είναι μια περιοχή με πολλά θέματα τεχνικά και άλλα που μπορούν να συζητηθούν. Ως εκ τούτου η διαχείριση είναι αρκετά περίπλοκη διότι εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις ε, ε, τεχνικές ομάδες, ομάδες δράσης όπως αποκαλούνται, έχουμε τη Γενική Συνέλευση, ε, είναι το ανώτατο επίπεδο εκπροσώπησης και εκεί κατά κάποιον τρόπο προκύπτει ένα πολύ σημαντικό σημαντικό παράθυρο για τις ε, μακροπεριφέρειες. Αν θέλετε αυτό είναι ένα παράθυρο μέσα από το οποίο γίνονται κάποιες φορές ε, πολιτικές ε, τοποθετήσεις που δεν γίνονται αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν φτάνουν στις ομάδες δράσης. Ως εκ τούτου, αυτό που μάθαμε, αν και είναι ίσως λιγάκι νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα, το βασικό μάθημα ε, είναι το εξής. Ε. Βέβαια αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Συνήθως δεν τα λέει αυτά δυνατά, αλλά το γεγονός ότι έχουμε ένα αυτόνομο, μια αυτόνομη μορφή ε, διαχείρισης δεν υπάρχει πολιτική δήλωση που να προκύπτει από την τεχνική συνεργασία. Ως εκ τούτου νομίζω ότι οι δύο αυτές περιοχές πρέπει να είναι αυτόνομες αλλά παρόλα αυτά ε, πρέπει να παρουσιάζουν και κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κατά την άποψή μου υπάρχει κάποια καθυστέρηση όσον αφορά τις ομάδες δράσης. Δεν έχουν επιτύχει ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή η Βαβαρία έχει την Προεδρία και προσπαθεί να ξεπεράσει τα προβλήματα παρουσιάζοντας τα δικά της τα ε, εμβληματικά προγράμματα που όμως δεν τα δέχονται άλλες ε, χώρες. Ε, αυτό δεν τη χάνει αναγνώρισης και ως εκ τούτου υπάρχουν αρκετές ε, ομάδες, ε, έχουμε τους φίλους των Άλπαιων, τους φίλους των ΜΕΝ, τους φίλους των ΔΕ, πάρα πολλούς φίλους ε, ε, και δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί τελικά, μπορεί να περνάνε προς το χρόνο στα μπαρ και στα εστιατόρια από το να κάνουν δουλειά. Συγγνώμη βέβαια για το στιάκι, που σας είπα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ομάδες αυτές αναγνωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια ότι Υπάρχει κάποιο περιθώριο για περιφερειακή και κεντρική συνεργασία και ε, συντονισμό. Οι τεχνικές πρωτοβουλίες προέρχονται από την βάση. Υπάρχει περιθώριο για διαφορετικές ε, θέσεις και απόψεις. Υπάρχει δυνατότητα να ε, αναζητηθεί ισορροπία και μετά να αρχίσει ο διάλογος σε τεχνικό επίπεδο. Υπάρχει και το πολιτικό επίπεδο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι πολιτικοί βέβαια μπορούν να ε, λένε αυτό που επιθυμούν γιατί προφανώς και γι' αυτό εξελέγησαν. Αλλά εγώ θα ήθελα να ισχυριστώ ότι το τελευταίο φόρουμ στο οποίο είχαμε τη συμμετοχή ε, κάποιων ε, εκπροσωπών αυτή δεν ήταν εθνικοί εκπρόσωποι, έγιναν κάποιες ε, δηλώσεις, αλλά δεν είχαμε άμεσα αποτελέσματα. Ίσως αυτά να προκύψουν στο μέλλον. Ας δούμε λοιπόν το μάθημα από όλα αυτά μέλλον. Και εδώ επιβεβαιώνω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοί μου, αλλά θέλω να κάνω και κάποια διαφοροποίηση. Αυτή η μακροπεριφερειακή συνεργασία είναι μια πολύ θετική εμπειρία. Χώρες, περιφέρειες, περιφέρειες ε, μιας ε, χώρας συναντιόνται Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπορεί κανείς και να ξεπεράσει ε, κάποιους στίχους, κάποια όρια. Όρια που να αφορούν σε ευρωπαϊκούς κανόνες και πολιτικές. Έχουμε λοιπόν στρατηγικές πολιτικές που αυτές έχουν σημασία για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάμε πέρα από την απλή συμμόρφωση. Αυτό μπορούν να συζητήσουν οι μακροπεριφέρειες. Κάθε φορά που καλούμε να συζητήσω πιθανές λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα, ε, είμαι αναγκασμένος ε, να ε, έρθω αντιμέτωπος με διάφορα διαρθρωτικά ταμεία, με διαφορετικούς κανόνες για τις διάφορες χώρες, διάφορους στόχους. Αυτό που θα έκανα στην Ιταλία είναι διαφορετικό με αυτό που γίνεται στην Σλοβενία. Όλα αυτά είναι λιγάκι απλουστευτικά. Και τέλος, θέλω να πω ότι υπάρχει και κάτι, ε, μια λέξη που θέλω να χρησιμοποιήσω, δεν υπάρχει ομοιογένεια, ε, ομοιογένεια των εργαλείων. Ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ισχυρός. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό τεχνικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή και επίσης να πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αν υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, τότε αυτό θα πρέπει να είναι ο πολιτικός φορέας για να συζητηθούν ορισμένα πράγματα. Και ε, θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει διάλογος και με τις αυτόνομες τεχνικές ε, ομάδες ε, οι οποίες προσφέρουν τεχνικές εξέλιξεις. να υπάρχει κεντρική και περιφερειακή εκπροσώπηση στο Συμβούλιο και στις ομάδες δράσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και η αυτονομία των ε, τεχνικών ομάδων. Και παράλληλα η διαχείριση ε, που πρέπει να έχει το Συμβούλιο για να καθορίζεται και το δρόμος που θα ακολουθηθεί. Τα πιο σημαντικά λοιπόν αποτελέσματα είναι όπως σας είπα να έχουμε την ευθυγράμμιση με τους κανόνες, με τους ε, φορείς, την ε, απλούστευση των διαδικασιών ε, χρηματοδότησης, έτσι ώστε να υπάρχει ευθυγραμμισμός, ευθυγράμμιση μάλλον με με τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επ' αυτού η Ιταλική θέση η θέση της αλληλικής κυβέρνηση είναι να προάγει τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, γιατί πράγματι υπάρχουν θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται σε μακροπεριφερειακό επίπεδο. Έχουμε την περιοχή του Δούναβη, της Άλπης, ε, τη Μεσόγειο διαφορετικές ε, περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε τον, ε, την απλούστευση των κανόνων για τις ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές, όπως επίσης και απλούστευση των κανόνων που διέπουν τους οργανισμούς αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μεγάλος ο κατάλογος των ομιλητών και προστίθενται και άλλοι συνάδελφοι. Ο κύριος Κουτσουρίνο πρώτος, που είναι ο εισηγητής μας ε, για την έκθεση εφαρμογής των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Ναι, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Ε, ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά δεν πάει καλά. Θα ήθελα να πω κάτι ουσιαστικό το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέξουμε και χάρη στα όσα μας λέτε εσείς ε, για τη συγκεκριμένη εμπειρία που ζείτε επί τόπου, που μου φαίνεται και ότι είναι και το πιο ενδιαφέρον. Εσείς μας ζητάτε να προωθήσουμε, να υποστηρίξουμε αυτή την πολιτική, να την εφαρμόσουμε και να την ε, προχωρήσουμε περαιτέρω. Η ουσία βέβαια είναι να δούμε πού θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Στα πλαίσια μιας αναθεώρησης της πολιτικής συνεχής της επόμενης ε, μήνες και φυσικά του δημοσιονομικού προ... Ε, των πολιτών των δημοσιονομικών προοπτικών τις οποίες θα συζητήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτρέψω ε, και βάσει και των όσων μας είπατε σήμερα το πρωί να μας υποδείξετε λίγο κάποια πράγματα βάσει και της εμπειρίας σας. Να μας πείτε δηλαδή για να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και μια νέα εποχή, η οποία θα πάει πέραν της πραγματικής δράσης και θα δώσει σε αυτή την μακροπεριφερειακή στρατηγική μια πιο συγκεκριμένη διάσταση ευρωπαϊκής πολιτικής. Να πάμε πέραν δηλαδή ε, του πειραματισμού. Αυτά τα οποία ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικά, σας τα αναφέρω εδώ επιγραμματικά, καταρχάς το πολιτές οικονομικό πλαίσιο. Μας λέτε ότι υπάρχει έλλειψη πόρων και, και ανθρωπίνου δυναμικού. Ωραία. Τι προτείνετε αρκεί ε, να ε, κάνουμε μια επίκληση στον ε, κανονισμό για την πολιτική συνοχή για το πλαίσιο 2014-2020. Πρέπει να πάμε παραπέρα υπό ποια μορφή και με ποιες προϋποθέσεις. Δεύτερον, κίνητρα, ε, κυρίως πολιτική διάσταση. Αυτό αφορά αποκλειστικά τις χώρες μέλη ή πρέπει να σταθούμε περισσότερο και στις περιφέρειες και το ρόλο των περιφερειών. Και αν αυτός ο ρόλος των περιφερειών δημιουργεί μεγαλύτερο ε, φόρτο, ε, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη δουλειά για τα κράτη-μέλη, κάπου λίγο δηλαδή να βρούμε ποια είναι η λύση και ποια είναι η διάμεση οδός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι ξέρω, βλέπω και το έγγραφο τώρα της Επιτροπής των Περιφερειών και θα δούμε και πώς θα πάει η έκθεσή μας, θεωρούν ότι στις μακροπεριφέρειες έχουμε μια δυνατότητα ε, να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις ε, ε, που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα. Και, για παράδειγμα, το μέσω ευελιξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κρίσεις αυτή τη στιγμή, κυρίως τη μεταναστευτική κρίση, τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την περιβαλλοντική κρίση, Μπορούν δηλαδή οι μακροπεριφέρειες να είναι υποψήφιες για να είναι ένα από τα πιθανά μέσα να βοηθήσουν την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Και αν ναι, με ποιο τρόπο. Θέτω απλώ ερωτήσεις. Τέταρτον, κάνουμε αναθεώρηση αυτή τη στιγμή της πολιτικής συνοχής. Ε, τι προτάσεις ε, μπορείτε να κάνετε από αυτού. Τι πρέπει να κάνουμε. Πώς ε, μπορούμε και στην αναθεώρηση του βασικού κανονισμού της πολιτικής συνοχής ε, για το διάστημα 2020-2027, τι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε για να μην είμαστε πλέον στο στάδιο του πειραματισμού, αλλά να είναι πιο ε, σωστά εφαρμοσμένη η πολιτική των μικροπεριφερειών. Και τέλος υπάρχει αυτό το αέναο θέμα της απλούστευσης, ένα θέμα το οποίο θίξατε όλοι σας. Αν ε, κατάλαβα καλά, κυρίως σας ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Ε, πρώτον οι διαδικασίες ε, αλλά και η διακυβέρνηση. Για αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να μας πείτε βάσει και της εμπειρίας σας σε ποια στοιχεία θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να ξεκινήσουμε κάτι. Εχθές ολοκληρώθηκε και η ομάδα εργασίας για την απλούστευση η Επίτροπος Τάισον και η Επίτροπο Σκρέτσο έκαναν και μία συνέντευξη τύπου και ξεκίνησαν αυτή τη συζήτηση βάσει και ε, τεκμηριωμένων κειμένων για την απλούστευση, αλλά το θέμα είναι ε, πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε εμείς, στη διακυβέρνηση ή στις διαδικασίες περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα ερωτηματικά, ε, τα οποία ήθελα να θέσω, γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσαν να διευκολύνουν και την ίδια μου την έκθεση. Να μην επαναλάβουμε με στήρο τρόπο αυτά που λέει η Επιτροπή των Περιφερειών, η πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου, η πρόσφατη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Να κάνουμε μια απόπειρα δηλαδή εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε κάποιε πιο συγκεκριμένε υποδείξει. Τι πρέπει να γίνει, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω ε, αναθεώρηση τη πολιτική συνοχή και ε, των πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το τώρα, τώρα στους σκιώδεις ε, εισηγητές. Ε, ο κύριος Μπόγκοβιτς έχει το λόγο πρώτα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και διαπιστώνουμε ότι το εργαλείο αυτό είναι αποτελεσματικό παντού ε, στην Σλοβενία. Εμείς συμμετέχουμε σε τρεις ε, μακροπεριφέρειες, στην ε, Αντριατική, Ιόνιο, αλλά και στις άλλες πρωτοβουλίες. Συμμετέχουμε σε όλες. Αυτά που ακούσαμε σήμερα ήταν πάρα πολύ καλά και ενδιαφέροντα και θέλω να ευχαριστήσω γιατί για μας ε, πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία μας προσφέρει την δυνατότητα να σκεπτούμε για το μέλλον της στρατηγικής. Εγώ θα μιλήσω για τη στρατηγική Αδριατική Ιόνιο. Αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Έχουμε δηλαδή τέσσερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερα εκτός. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή μπορεί κανείς να δει πολύ συγκεκριμένα πώς λειτουργεί η συνεργασία ανάμεσα σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτα κράτη. Και επίσης συνεργασία ανάμεσα σε κράτη που κατά το παρελθόν είχαν μεγάλα προβλήματα. Ξέρετε γιατί, λόγω των γεγονότων στη Γεγκοσλαβία τη δεκαετία του 90. Αυτή λοιπόν η μυσαλλοδοξία και τα προβλήματα που υπήρχαν κατά το παρελθόν σε κάποιο βαθμό εξακολουθούν να υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που διακυβεύεται είναι το οικονομικό. Πρόκειται κυρίως για θέματα συνεργασίας, τον τουρισμό και σε αντίθεση με τις ε, χώρες Ανατολικής Ευρώπης, ε, για μας η βάση συνεργασίας αρχικά ήταν πολύ χειρότερη και νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιες ε, δυσκολίες όσον αφορά το μελλοντικό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να τις ε, παραμελήσουμε αυτές τις μακροπεριφέρειες. Ε, πρέπει οι περιφέρειες αυτές να παίρνουν κονδύλια και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι για τους στόχους των μακροπεριφερειών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και εθνικοί και περιφερειακοί προϋπολογισμοί και πρέπει επίσης να ε, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία σε κονδύλια που όπως σας είπα έρχονται από διαρθρωτικά ταμεία, από το Ταμείο των Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ δηλαδή, ε, κονδύλια από το πρόγραμμα Horizon, από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορέσουμε ε, να ενισχύσουμε αυτό το αίσθημα του ανήκειν σε αυτές τις περιφέρειες. Κυρίως μιλάω για αυτή που μιλάω εγώ, για την περιφέρεια των Άλπαιων. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ορισμένα πράγματα, ευχαριστώντας όλους όσους πήραν το λόγο πριν από μένα. Θα ήθελα να πω, ε, κατ' ουσίαν, ότι συμφωνώ με όλα όσα είπαν. Νομίζω ότι η προσέγγιση που ακολούθησαν ε, ήταν καταρχάς αναλυτική. Εγώ πάντως από πλευράς μου δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτήν την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ε, ε, ε, ακολουθούμε μια προσέγγιση κάπως πειραματική. Με την εξαίρεση της Βαλτικής θάλασσας πιστεύω ότι όλη η διαδικασία και η περιγραφή αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά προσπαθεί να ξανακολλήσει τα κομμάτια της αποτελεσματικής Ευρώπης που έχουν διασπαρεί από εδώ και από εκεί. Εγώ θυμάμαι το 2005 όταν δημιουργήθηκε αυτή η περιοχή, η περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιωνίου. Ε, ήμουν δήμαρχος τότε και θυμάμαι την κατάσταση. Καταλαβαίνω πολύ καλά τα τρία όχι τα οποία εμφανίστηκαν όταν, άρχισαν, ε, όταν αρχίσαμε να συζητούμε τη στρατηγική. Αυτέ οι τρει αρνήσεις όμω δεν, ε, δεν έχουν καλή ε, βάση. Πρέπει να σκεφτούμε μία δομή συντονισμού που θα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Εγώ σκέφτομαι την περίοδο, την περιφέρεια συγγνώμη, της Αδριατικής και τους δήμους και τις πόλεις που μπορούν να συμμετέχουν. Συμμετέχουν λίγο τελικά, γιατί ε, ε, τα κράτη-μέλη ενδεχομένως να ενδιαφέρονται λιγότερο από τους δήμους και τις πόλεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια δομή πιο ισχυρή γιατί διαφορετικά θα υπάρξει ένας κατακαιρματισμός μέσα στο χάος που δεν θα επιφέρει τίποτε. Επίσης, πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το όλο θέμα. Ας είμαστε συγκεκριμένοι. Έχουμε προγράμματα συνεργασίας Ιταλίας, Κροατίας, Ιταλίας, Σλοβενίας, Σλοβενίας, Κροατίας, ε, πρόγραμμα με την Αλβανία, με το Μαυροβούνιο, με τη Σερβία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πολύ καλά είναι, όλα αυτά έχουν προέλθει από το παρελθόν, από την πολιτική συνοχή, αλλά μήπως θα μπορούσαμε και εδώ να αναζητήσουμε μία λύση που θα μας επέτρεπε να αλλάξουμε λίγο την κατάσταση, γιατί εγώ είμαι ένας ε, από εκείνους ε, που κατάφεραν την εφαρμογή πολλών τέτοιων προγραμμάτων και δεκάδες εκατομμύρια έχουν ε, δαπανηθεί όχι πάντοτε με το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Βέβαια, πολλοί κόσμοι ήταν ικανοποιημένος, δεν λέω το αντίθετο, αλλά δεν πρέπει να σταματούν τα πράγματα εκεί. Πρέπει να αναζητούμε έναν τρόπο αντιμετώπισης όλων αυτών των διμερών προγραμμάτων που υπάρχουν ήδη, έναν καλύτερο τρόπο. Αν θέλουμε να καταστεί αποτελεσματική μια μακροπεριφερειακή στρατηγική, πρέπει να δούμε μια βάση χρηματοδότηση στρατηγικών αυτών και των προτεραιοτήτων που θα καθοριστούν μεταξύ των ε, κρατών μελών που ε, συμμετέχουν. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτό που αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ε, μακροπεριφέρειας Αδριατικής Ιωνίου. Νομίζω ότι θα ήταν πιο αποτε... Θα, θα, πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην ανταπόκριση σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών μας, η κυρία ε, θα ήθελα να, στείλω ένα γράμμα στην κυρία κρέντσου, η οποία θα έλεγε, το οποίο θα έλεγε ότι οι πόλεις ε, της περιφέρειας Αδριατικής Ιωνίου ε, συμφώνησαν όλες γύρω από μία σειρά πρωτοβουλειών και ζητούν από την Επίτροπο να προαχθεί κάτι τέτοιο. Και νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι έχει φτάσει πλέον η χρονική στιγμή να βγούμε από αυτή την πειραματική προσέγγιση και να περάσουμε σε μια πραγματική φάση εφαρμογή. Γιατί οι συμπολίτε μα που ζουν στο έδαφο αυτών των μακροπεριφερειών περιμένουν από εμά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κύριε κύριο Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι οι σημερινέ παρουσιάσει από τους ειδικού που έχουν και την εμπειρία της εφαρμογής μας βοηθούν να επιχειρήσουμε αυτό που μόλις ανέφερε πριν από λίγο ο κύριος Κοζολίνο. Να μην κάνουμε μία έκθεση ρουτίνας, αλλά να δούμε με τη συμβολή και της εμπειρίας από τη μέχρι τώρα εφαρμογής και της θετικής εμπειρίας και των δυσκολιών, πώς αυτή η συνεργασία στις μακροπεριφέρειες θα γίνει πιο αποτελεσματική, πιο χρήσιμη για τους πολίτες με πιο ορατά αποτελέσματα. Ε, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ε, σε μία από τις τοποθετήσεις των ειδικών από τον πρώτο μιλητή, ότι δεν μιλάμε απλώς για μια συνεργασία ανάμεσα σε κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να έχουν μια προοπτική ένταξη. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό που αφορά την αξιοποίηση από κοινού σε προγράμματα για τις μεταφορές, την ενέργεια, συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, όπου η κλίμακα της μακροπεριφέρειας επιτρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μιλάμε για μια αντίληψη που βοηθάει με την κλίμακα της μακροπεριφέρειας να κάνουμε πράγματα που ο καθένας μόνος του δεν μπορεί. Όταν μιλούμε για πόλεις, για περιφέρειες και αυτό απαιτεί μια ε, διαφορετική ε, προσέγγιση. Εγώ θα ήθελα ε, να επισημάνω και κάτι ακόμη. Έχουμε δύο μακροπεριφέρειες που έχουν προχωρήσει περισσότερο και έχουν εμπειρίες στη Βαλτική και στο Δούναβι και άλλες δυο οι οποίες είναι πιο πίσω γιατί ξεκίνησαν αργότερα. Ειδικά για αυτήν που αφορά και στη χώρα μου την Ελλάδα, Αδριατική Ιόνιο και έχουμε και την πρόσθετη δυσκολία που ήδη αναφέρθηκε ότι μιλάμε για χώρες, τέσσερις μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέσσερις μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πριν λίγα χρόνια είχαν πολεμικές αντιπαραθέσεις μεταξύ τους κάποιες από αυτές. Και υπάρχουν και μεγάλες, μακραίωνες ε, αντιθέσεις. Άρα θα έλεγα ότι το πρώτο που πρέπει να διασφαλίσουμε μέσα από αυτή την έκθεση ή δυνατόν με την ευρύτατη δυνατή συνένεση και συμφωνία είναι ότι οι μακροπεριφέρειες πρέπει να προχωρήσουν να μην οχυρωθεί κάποιος τεχνοκράτης στις Βρυξέλλες πίσω από υπαρκτά προβλήματα και δυσκολίες και να πει επειδή τώρα θα λιγοστέψουν και τα χρήματα να τις υποβαθμίσουμε αυτές τις στρατηγικές επιλογές. Χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση από τις Βρυξέλλες και όχι λιγότερη. Το δεύτερο είναι ότι τα κονδύλια, επειδή ανήκει και μια συζήτηση για τις πολιτικές συνοχής και μετά το 2020. Τα κονδύλια για αυτή την επιλογή τη συνεργασία σε επίπεδο μακροπεριφερειών δεν πρέπει να μειωθούν. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίξει στεναρά η Επιτροπή Περιφερειών. Και τα κονδύλια που δίνονται από τις πολιτικές συνοχής, που είναι τα περισσότερα, και τα κονδύλια που δίνονται από κεντρικότερα κομμάτια του κοινοτικού προϋπολογισμού, όπως είναι το Horizon. Δεν πρέπει. Αντίθετα πρέπει να δώσουμε βάρος σε πρακτικές ιδέες και προτάσεις στηριγμένες στην εμπειρία για το πώς μπορεί να γίνει πιο μετρήσιμο το αποτέλεσμα για τον πολίτη και την κάθε περιφέρεια. Και εκεί νομίζω ότι η λέξη κλειδί που ήδη ακούστηκε είναι απλούστευση και μεγαλύτερη προβολή των όποιων θετικών βημάτων έτσι ώστε να πιστούν περισσότερο οι περιφέρειες, τα κράτη-μέλη το πολιτικό επίπεδο ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με αυτό το θέμα. Γιατί έχουμε, δεν έχουμε πάντα από, την πολιτική, ε, από το πολιτικό επίπεδο την επαρκή ε, ε, ανταπόκριση. Το δεύτερο, το τεχνικό επίπεδο είναι πολύ διαφορετικό, σωστά υπόθηκε από, τους, από κάποιον από τους ειδικού και καμιά φορά ε, η πολιτική δεν στηρίζεται στα τεχνικά δεδομένα, προσπαθεί να τα υπερκεράσει και έτσι δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Το τελευταίο που θέλω να πω. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στην αποδοτική συνεργασία των θεσμικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιοχή, για παράδειγμα, της Αδριατικής Ιωνίου ασχολούνται κι άλλοι, διάφορα λόμπις. Ε, όπως είπε ο, ο Ιταλός καλά είναι αυτά, αλλά δεν είναι η δουλειά μας να υποκαταστήσουμε τις θεσμικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δουλειά των λόμπις. Και επειδή καμιά φορά αυτά τα πράγματα αναφέρονται και μπαίνουν στο ίδιο καλάθι, νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε στην έκθεση που θα ετοιμάσουμε ότι εμάς μας ενδιαφέρει η στρατηγική επιλογή των μακροπεριφερειών να ενισχυθεί μέσα από τα θεσμικά εργαλεία που υπάρχουν και όχι και από παράπλευρες επιλογές που επιρετούν ενδεχομένως και γεωπολιτικές επιδιώξεις ορισμένων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρλετς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πιστεύω οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι πολύ σημαντικές ε, όπως όμως είπε ήδη ο συνάδελφος κύριος Γιάκοφ έχουμε την τάση να τα περιορίζουμε όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό σε, ε, στο επίπεδο του πειραματισμού, το βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι στρατηγικές, πώς ε, διατίθεται τα κονδύλια, τα κονδύλια και πώς ε, γίνεται η εφαρμογή. Νομίζω ότι σε μερικέ περιπτώσει, έχουμε πολλέ φορέ πει ότι τα, τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τι στρατηγικέ και βλέπουμε τέτοιου είδου προβλήματα σε υψηλότερο επίπεδο τη πολιτική ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε στι συζητήσει ε, ε, και τι διαθεσμικέ, τι διοργανικέ, Σκέφτομαι για παράδειγμα το θέμα του ενεργειακού πακέτου. Μιλάμε και σε αυτήν την περίπτωση για μια περιφερειακή προσέγγιση, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, φέρεται ως ε, εκείνη που προωθεί αυτήν την προσέγγιση ε, δεν έχει υποστηρίξει επαρκώς την μακροπεριφερειακή στρατηγική και την πρόοδό της. Ένα τμήμα των προτάσεων και των συστάσεών μας θα έπρεπε συνεπώς να εστιάζει στην ε, ενίσχυση των μακροπεριφερειακών ε, στρατηγικών και στο να προωθούνται ε, σύμφωνα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό προγραμματίζεται όσοι έχουν ε, μια, μια εμπειρία από διακυβέρνηση πειραματική που βασίζεται σε καλή θέληση, ε, θα ξέρουν ότι έχει σημασία να περάσουμε σε μια πραγματική διαδικασία λήψης αποφάσεων που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν να συμφωνήσουν επί των στρατηγικών ε, και των στόχων και επίσης πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένα όργανα τα οποία θα είναι πλήρως υπεύθυνα στο πλαίσιο των περιφερειών για τη διαχείριση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ των ε, πολιτικών και της, του καθορισμού τους για την περίοδο μετά το 2020 όταν μιλάμε για τις μεταφορές, την διασύνδεση, την ενέργεια πρόκειται για τομείς που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για για την επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο και πρέπει συνεπώ να ενσωματωθούν στην μακροπεριφερειακή στρατηγική. Γι' αυτό πιστεύω ότι η διακυβέρνηση των ε, μακροπεριφερειών αυτών πρέπει να βελτιωθεί ώστε να εξασφαλίζεται μια καλή, μια ορθή διαχείριση των σχετικών κονδυλίων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταμάτου, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ρεαλίστια ε, δυστυχώ και να σα ζητήσω να είστε κι εσεί ρεαλιστέ. Συμφωνώ μεν ότι το θέμα της στήριξη ακόμα και της χρηματοοικονομικής είναι θεμελιώδη σημασία, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, ότι θα υπάρξουν ε, ε, μελλοντικέ περικοπές κυρίως στην κοινή γεωργική πολιτική και στην πολιτική συνοχή. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε οικονομική στήριξη για τις μακροπεριφέρειες. Πέραν αυτού, έστω ότι είναι δυνατό, εμείς ε, από πλευράς μας ως ευρωβουλευτές θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη θέση με περισσότερα στοιχεία για την επίδοση των μακροπεριφοριών πόση ανάπτυξη, πόση απασχόληση ε, έχουν δημιουργήσει μέχρι τώρα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσουμε τώρα τον κατάλογο των ε, ομιλητών. Ευχαριστούμε κύριε Νταμάτο, κύριο Νίλσεν. Ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι μια νέα πτυχή και συνεπώς πρέπει να οργανωθεί μια παρακολούθησή τους, να δούμε κατά πόσο χρειάζονται τροποποιήσεις. Η δική μου εμπειρία βασίζεται στη Σουηδία και στην ε, μακροπεριφέρεια της Βαλτικής. Εγώ πραγματικά συμμετείχα σε μεγάλο βαθμό σε τοπικό επίπεδο όταν ξεκίνησε αυτή η δουλειά και όλα όσα άκουσα ενισχύουν την ε, δική μου αίσθηση και τη δική μου εμπειρία ότι δεν υπάρχει δηλαδή οικειοποίηση αυτών των στρατηγικών. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε τα κράτη-μέλη όμως, ε, ούτε οι, τα όργανα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Οι περιφέρειες αντιθέτως είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές, πολύ δραστήριες, έχουν προσπαθήσει να συνεργαστούν. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος είναι ο κατάλληλος ρόλος ε, των ε, μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχουν ε, μίνι ευρωπαϊκές ενώσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λέω ότι όταν μιλάμε για ένα ισχυρό σύστημα, δεν εννοούμε ότι πρέπει να, να διαιρέσουμε την Ευρώπη σε πολλές μικρές ευρωπαϊκές ενώσεις, όμως, από τη μία πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και πιστεύω ότι θα έπρεπε να περιοριστούμε στους τομείς ε, επί των οποίων τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλη αρμοδιότητα όπως η θαλάσσια πολιτική, η περιβαλλοντική πολιτική, ε, σκέφτομαι επίσης και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πρέπει επίσης να δούμε όλη αυτή την προσπάθεια ως τρόπο ενίσχυσης της ε, διασυνοριακής συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω ότι στην πολιτική συνοχή θα είναι εύκολο να βρούμε τα εργαλεία για να οργανώσουμε αυτήν την ενίσχυση στην αρχή 5% των περιφερειακών κονδυλίων ε, ήταν δεσμευμένα για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Δηλαδή οι περιφέρειες έπρεπε να βρουν εταίρους σε άλλες χώρες Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται νέα ε, πρικοδότηση από τον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε πού θα πάνε τα συγκεκριμένα κονδύλια, λέγοντας ας πούμε τόσο τις 100 πρέπει να ε, πηγαίνει στην μακροπεριφερειακή στρατηγική. Αυτό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να δημιουργηθεί καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Για μένα, σε τελική ανάλυση, Το βασικό είναι να υπάρξει αυξημένη συνεργασία μεταξύ των, των περιφερειών σε διασυνοριακό επίπεδο, ε, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανάκαμψης, ε, πολιτισμικής ανάπτυξης και επίσης οικοδόμησης ε, της Ευρώπης κάπως πιο ειρηνικής. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και σε όσους και στους προσκεκλημένους μας, ομιλητές μας, αλλά και στους συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή ε, σχεδιάζεται το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας αφορά ακριβώς αυτό. Η, έμφαση ε, λέγεται ότι θα, έπρεπε, θα, θα, θα δοθεί στο να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους. Η βασική πρόκληση λοιπόν για τις μακροπεριφέρειες ε, είναι να έχουν τα προγράμματα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Το βασικό επιχείρημα λοιπόν που θα έπρεπε να ε, θέσουν οι, οι μακροπεριφέρειες είναι ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής και της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών μπορεί να υπάρξει περισσότερη προστιθέμενη αξία για την επίτευξη, προς την επίτευξη των κοινών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα την εξάλληψη των αποκλεισμών, την μπλε ε, οικονομία. Ε, νομίζω ότι υπάρχει υπάρχουν πόροι που δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς και αυτή είναι η, η κοινή ταυτότητα που μοιράζονται οι περιφέρειες που απαρτίζουν τη μακροπεριφέρεια. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν ε, στις ετήσιες συναντήσεις 700-800 εμπλεκομένων φορέων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι πρακτικοί, είναι επιχειρηματίες, ε, είναι από τοπικές ε, αρχές, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αν χρησιμοποιηθεί και ενισχυθεί αυτό το δυναμικό με το σωστό τρόπο, πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό που είπε ο κύριος Νίλσεν, δηλαδή ένα ποσοστό ε, των κονδυλίων ε, να εφεθεί κατά μέρος προκειμένου να ε, μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η προστιθέμενη αξία της λειτουργίας των μακροπεριφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εδώ έναν πολύ συγκεκριμένο και ε, σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Όπως επίσης και οι ε, διαχειριστικοί φορείς ε, των μακροπεριφερειών. Το θέμα της απλούστευσης είναι επίσης σημαντικό, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάτι το οποίο υπόθηκε ήδη. Η το βασικό θέμα είναι οι στρατηγικές, οι μακροπεριφερειακές, να συμπεριληφθούν σε ευρύτερους στόχους Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ρόπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον ε, αυτά που ελέγχθησαν. Ε, ακούσαμε βέβαια ε, προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς αν θέλει να εφαρμόσει περιφερειακές στρατηγικές. Οφείλω να σας πω ότι εμείς ε, κατανοούμε πάρα πολύ καλά ότι τα προγράμματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και προφανώς ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, στο μέγιστο αυτές τις στρατηγικές. Παρουσιάστηκε και η εμπειρία της Λετωνίας και χαίρομαι πάρα πολύ που η περιοχή της Βαλτικής παρουσιάζεται σε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Φαντάζομαι όμως ε, θα ακούσατε επίσης ε, ότι η συμμετοχή δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό δεν ελέγχθη πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι οι στόχοι και οι προτεραιότητες να μην έχουν οριστεί με την ε, δέουσα ακρίβεια. Κατόπιν τούτου το θέμα αυτό δεν πρέπει να το θίγουμε μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο συνεργασίας εταίρων. Δηλαδή όλες αυτές τις ε, απόψεις πρέπει κάπως ε, να τις ε, επιλέξουμε και να τις διαμορφώσουμε με τέτοιο τρόπο που να οδηγούν σε κάτι το κοινό. Γιατί αν υπάρχει κοινή προσπάθεια, τα αποτελέσματα είναι και πολύ καλύτερα. Ας πάρουμε το παράδειγμα της ε, κλιματικής αλλαγής. Τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτό το τομέα θα μπορούσαν παραδείγματο χάρη να είναι ε, προτεραιότητα τουλάχιστον ε, για την περιοχή της Βαλτικής. Για μας αυτό θα μπορούσε να είναι άλλη μία προτεραιότητα, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν, δηλαδή η ενέργεια και όλες οι άλλες. Και με τον τρόπο αυτό ε, θα μπορούσαμε να ε, δημιουργήσουμε μία γέφυρα προς ε, τα μέτρα που λαμβάνονται για την κλιματική αλλαγή. Σήμερα γίνεται λόγος για την απλούστευση. Το πρόγραμμα Omnibus είναι ένα πρόγραμμα που συζητείται ευρέως και φαντάζομαι ότι περιμένετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Εμείς ελπίζουμε στο πλαίσιο της ε, συνοχής ε, να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα η προοπτική μετά το 2020, η κατάσταση μετά το Brexit. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οφείλουμε να καταβάλουμε προσπάθειες από κοινού για να επιτύχουμε στόχους που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση, όταν δηλαδή θα περιοριστούν τα κονδύλια. Η συνεργασία δεν θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με, μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλη να είναι η εξέλιξη. Διότι το κύριο καθήκον είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί. Κυρία Τόμασιτς, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ορισμένα πράγματα. Εγώ είμαι από την Κροατία και προφανώς άκουσα με πολύ προσοχή την στρατηγική για την Αδριατική και ε, το Ιόνιο. Συγκράτησα κάποια προβλήματα, τα οποία, αν κατάλαβα καλά, είναι τα βασικά προβλήματα. Δεν έχω ερωτήσεις προς τους ομιλητές, προς τους προσκεκλημένους μας. Έχω κυρίως ερωτήματα να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν προβλήματα με την διοικητική ικανότητα. Δεν υπάρχει αρκετή ε, αρκετά σωστή διαχείριση ε, που να οδηγεί στη σωστή εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Θα ήθελα να μάθω η Επιτροπή τι προτείνει για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοδότηση με πιο αποτελεσματικό τρόπο και σε ποιο βαθμό ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα της τεχνικής αρρωγής για να ενισχύσουμε τη διοικητική ικανότητα των κρατών μελών και την ενίσχυση συνεπώς ε, της, ε, της ε, μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο. Πρέπει και οι, και οι πολίτες να συμμετέχουν. Σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν ενεργά στο πλαίσιο αυτής της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Η κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ στην αίθουσα ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει να συνεχιστεί και θα σας εξηγήσω και γιατί. Συμφωνώ βεβαίως με τον κύριο Παπαδημούλη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Πώς μπορούμε όμως να συνεχίσουμε και μάλιστα ε, να πάμε και πέραν αυτών, όπως είπε κάποιος από τους προλαλήσαντες. Θα ήθελα να πω δύο λόγια ως ε, μέλος του Κοινοβουλίου που συμμετείχε σε δύο από τις αιτήσεις συνεδριάσεις της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής στην Κροατία και στην Ελλάδα. Και να ξεκινήσω με το τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Χρειάζεται ε, πράγματι ένα ακόμα χρηματοδοτικό μέσο για να χρηματοδοτήσουμε τις μακροπεριφέρειες. Κατά την άποψή μου όχι αρκεί να προχωρήσουμε με συμπληρωματικό τρόπο, να συνεχίσουμε με την προσθετικότητα, τη συμπληρωματικότητα, αλλά όχι με ένα επιπλέον μέσο, με έναν ακόμα κωδικό στις πολιτικές δημοσιονομικές προπτικές. Και επίσης πρέπει να ζητήσουμε τεχνική συνδρομή. Γι' αυτό και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Δεύτερον, η τα δέλεαρ των μακροπεριφερειών. Είναι δελεαστική μακροπεριφέρεια. Κατά την άποψή μου, όχι αρκετά. Δεν απευθύνεται αρκετά στις πόλεις, στις περιφέρειες, ούτε καν στα κράτη-μέλη. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν είναι απλούστερο, δεν είναι δελεαστικό και δεν προσφέρει κάτι το οποίο να οδηγεί σε αποτελέσματα. Και ε, με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω και την σύντομη παρέμβασή μου. Θα ήθελα να ζητήσω μια έκθεση για την εφαρμογή από τους συμμετέχοντες, ε, όχι από εμά, από αυτούς που συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα. Ε, πρέπει να δούμε δηλαδή πώς εφαρμόζονται επιτρόπου οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Και όπως ξέρετε η Ελλάδα συμμετέχει στη στρατηγική για την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής του Ιωνίου και θα ήθελα να ξέρω πόσοι συμμετείχαν ήδη σε αυτή τη στρατηγική και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και επίσης ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονες μας ε, που παρουσίασαν ε, τις ε, μέχρι τώρα καταβληθήσεις προσπάθειες για την μακροοικονομική συνεργασία. Πριν από 8 χρόνια η πρώτη μου δουλειά εδώ στο Κοινοβούλιο ήταν να αναλάβω σκιώδης ηγητής για την στρατηγική για τη Βαλτική. Πέρασαν 8 χρόνια και όσον αφορά την εφαρμογή μακροοικονομικών και μακροπεριφερειακών στρατηγικών, να σας πω κάτι, δεν έχουμε προχωρήσει και πολύ. Αρχικά, η μακροπεριφερειακή στρατηγική είχε ως στόχο να επιλέξει ένα συγκεκριμένο θέμα που να αφορά διάφορα κράτη-μέλη. Και μετά αυτά τα κράτη από κοινού και συμπεριλαμβάνοντας βέβαια και τους φορείς που υπήρχαν σε αυτές τις ε, χώρες και τις περιφέρειες να δεσμευτούν για ένα συγκεκριμένο στόχο. Στόχος ήταν τότε ε, το περιβάλλον. Η Βαλτική θάλασσα έχει ως παράκτης χώρες και χώρες ε, όπως η Ρωσία. Αυτή η Βαλτική θάλασσα επιβαίνεται πάρα πολύ από τις εισρωές στην ε, θάλασσα αυτή και όσον αφορά την ε, ε, επιβάρνηση... στην Βαλτική έχουμε πάρα πολλά σκάφη που τη διασχίζουν, άρα δηλαδή θα έπρεπε να τεθούν κάποιες προδιαγραφές για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα της εσωτερικής ναυσιπλοείας στην Βαλτική. Στην περίπτωση του Δουνάβεως εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αυτό που ενδιέφερε ήταν ο Δούναμπης να προβληθεί ως μια περιοχή που ε, μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη των κρατών της Βάδης Βιτεμβέργης, ε, της Αυστρίας, ε, να υπάρξουν περισσότερες, περισσότεροι οικονομικοί δεσμοί με, των χωρών αυτών με τα Βαλκάνια. Ως εκ τούτου ε, να υπάρχει κάποια οικονομική ζώνη από τη Βάδη Μιτεμπέργη μέχρι τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Όλα αυτά έχουν κάποιες δυνατότητες επιτυχίας μόνο εφόσον οικειοποιηθούν τα κράτη που τα, που τα αφορά η στρατηγική, τη στρατηγική αυτή. Ξέρετε κάτι, ε, υπάρχουν αρκετά εργαλεία, διαρθρωτικά, κονδύλια, ε, προγράμματα Interreg, αυτό που χρειάζεται είναι, όπως σας είπα, να οικειοποιηθεί κανεί ένα πρόγραμμα. Τι γίνεται όμως, βιώνουμε ότι όλες οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές μακροπεριφερειακής συνεργασίας, όλες οι χώρες ασχολούνται με άλλα θέματα. Παραδείγματο χάρη, από την Πολωνία έχουμε τώρα την πρόταση να δημιουργηθεί μια περιφέρεια που να αφορά τρεις θάλασσες, Βαλτική, Πόντο και Ανδριατική. Και λένε να συνεργαστούν αυτές οι τρεις θάλασσες, ε, να βρουν μια μορφή πολιτικής συνεργασίας ε, οι παραθαλάσσιες περιοχές. Μην ξεχνάτε, είχαμε και τις ε, χώρες Βίζεγκάρτ, οι οποίες βέβαια έχουν καθαρά πολιτικούς στόχους. Και σήμερα διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει τις έξι υποψήφιες χώρες των Βαλκανίων και γι' αυτό θα ε, υπογράψει διάφορα προγράμματα που θα ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση των χωρών αυτών. Στην Τριέστη θα έχουμε Αλβανία, ε, Μακεδονία, Μαυροβούνη, Σερβία, ε, με εκπροσώπους από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες δηλαδή, των Βαλκανίων θα συναντούν με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε τους ίδιους στόχους που υποτίθεται ακολουθεί η μακροπεριφέρεια του Δουνάβης. Τώρα τι είναι αυτό πάλι. Άλλη πρωτοβουλία καινούργια πρωτοβουλία. Μα τι γίνεται. Υπάρχει άραγε κάποια συνέπεια στους ε, μακροπεριφερειακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθορισμένο το ποιος κάνει τι, πώς κατανέμονται αρμοδιότητες. Και θεωρώ ότι ε, σήμερα από αυτά που λέξαμε πρέπει να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα και μακρά η συζήτηση. Και τώρα η πρόκληση είναι για τους ε, προσκεκλημένους μας. Θα πρέπει σε δύο λεπτά ο καθής να προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να μας πείτε και την άποψή σας ε, για τα όσα ακούστηκαν. Ποιος θα λάβει το λόγο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω πέντε πράγματα πολύ σύντομα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε είτε πειραματικά είτε ε, με πειραματίστικο τρόπο. Δεν έχει σημασία ο όρος. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε με κάποιο τρόπο τα πράγματα. Ε, και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι διαφορετικής ηλικίας. Έχουμε δύο ε, βρέφη και δύο που είναι σχεδόν στην εφηβεία. Πρέπει να τα αφήσουμε να προχωρήσουν γιατί είναι σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξη και δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Δεύτερον, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουν να χωρίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να είναι πρωτίστω Ευρωπαϊκέ Στρατηγικέ, να ε, εφαρμόσουν συνολικέ. Ε, πολιτικές Ευρωπαϊκές Ένωσης σε συγκεκριμένο ε, καθορισμένο χωρικό πλαίσιο. Και φυσικά μπορεί να παρέμβουν και άλλες πολιτικές, πολιτική διεύθυνση και ούτω καθεξής και να έχουμε διαφορετική σύνθεση από εκεί και πέρα. Και συμφωνώ ότι αυτό μπορεί να συγχύσει λίγο. Αλλά έτσι έχει πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και δεν μπορούμε να ε, περιμένουμε οι μακροπεριφέρειες να είναι ε, πιο αποδοτικές και να έχουν καλύτερη απόδοση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, νομίζω ότι υπάρχουν δύο επιλογές και είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υπάρχει ανάγκη για περικοπές, ε, δεν θα υπάρχουν περισσότερα χρήματα, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ακόμα και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές λοιπόν πρέπει να αναγνωριστούν σε εθνικά κάθετος ευρωπαϊκά συνολικά προγράμματα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο για τις μακροπεριφερειακές ε, στρατηγικές. 5% ακούστηκε, 10% δεν ξέρω. Αυτά είναι υποδιαπραγμάτευση. Η άλλη λύση θα ήταν να ε, έχουμε ε, κλασικά διεθνή προγράμματα, αλλά εδώ ελοχεύει πραγματικά ο κίνδυνος ε, να ξαναπέσουμε σε εδαφικά προγράμματα. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές δεν είναι μόνο εδαφικές στρατηγικές, είναι κάτι περισσότερο. Τέταρτον, σαφώς οι στρατηγικές πρέπει να είναι στρατηγικές, που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε τι έχουν λάβει υπόψη. Μπορεί να μην έχουμε πάρα πολλού στόχους όπως έχουμε τώρα, να πρέπει να περικόψουμε και να βρούμε ποια είναι τα εμβληματικά προγράμματα, όχι μόνο για την κάθε χώρα της μακροπεριφέρειας, αλλά για όλη την μακροπεριφέρεια. Και τέλος, κατ' εξίσου σημαντικό, δεν θα πρέπει να ξεναχνούμε και την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσεγγίσει και τα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε να υπάρχει και καλύτερη παρακολούθηση ε, σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι μπορείτε να τα καταφέρετε λοιπόν σε δύο λεπτά. Κυρία μου, παρακαλώ. Ναι, νομίζω και εγώ πέντε έχω να πω. Χρηματοδότηση πρώτα-πρώτα. Σε πολλές συζητήσεις εδώ ε, διαπιστώνουμε και λέμε πάντα ότι δεν υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση. Αλλά πρέπει να συντονίσουμε όλα αυτά τα μέσα χρηματοδότησης που έχουμε. Υπάρχει πολιτική συνοχή, υπάρχουν προγράμματα, το ορίζοντα 2020, το LIFE, το EFSI το Connecting Europe Facility. Υπάρχουν τόσα πολλά και διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, πρέπει απλώς να τα συντονίσουμε με καλύτερο τρόπο. Ε, Εχθέ στο αεροπλάνο σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να γίνει, πώς μπορούμε να τα συντονίσουμε όλα αυτά καλύτερα. Και σκέφτηκα το εξής. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει κάτι νέο για την διεθνική συνεργασία, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα προγράμματα που έχουμε, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Επίσης ε, πρέπει ε, στο μέλλον να μην βασιζόμαστε μόνο στην πολιτική συνοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε αφιερώσει πολλά στην πολιτική συνοχή. Ε, λέμε ότι είναι η μεγαλύτερη πολιτική της Ένωσης με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση. και οι άλλες ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές αλλά και η στρατηγική για το Δούναβι ε, χρηματοδοτείται κυρίως από την πολιτική συνοχή. Αλλά έχουμε και την πραγματικότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Μεταναστευτική κρίση, Brexit. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμίσουμε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει καλύτερο συντονισμός. Αν ή καθέν θεωρούσα ότι προσωπικά είμαι καλύτερη στην πρακτική εφαρμογή παρά στις ρητορίες. Και με όλο το σεβασμό προς τους πολιτικούς, νομίζω ότι το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν οι πολιτικοί είναι να μιλήσουν για αυτές τις στρατηγικές, για να αυξήσουν την προβολή τους. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να αυξήσουμε και τις δυνατότητές μας και τις ε, δεξιότητες αυτών που εφαρμόζουν αυτές τις ε, στρατηγικές. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις δεξιότητες ε, των ε, θεσμών και των οργάνων που ασχολούνται απευθείας με αυτούς που εφαρμόζουν τις στρατηγικές και τους project manager. Σήμερα άκουσα αρκετές φορές να αναφέρεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος των κρατών μελών και των περιφερειών που συμμετέχουν. Και τώρα διαπιστώνω ότι ε, με αυτό το παιχνιδάκι. Πάει το μπαλάκι από τον ένα στον άλλον. Κατά την άποψή μου λοιπόν, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρός εδώ, διότι η εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών βασίζεται σε πολύ περίπλοκα συστήματα. Διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικές διαδικασίες, αριθμός θεσμικών οργάνων ε, και άλλων αρμοδίων φορέων. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να είναι ισχνότερο σε μία περίπτωση, όταν υπάρχουν ε, τα προγράμματα πλέον, τα οποία θα προχωρούν από μόνα τους και δεν θα χρειάζεται εμείς να τα πιέσουμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Και ένα τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, ε, ακούστηκαν πολλά για την αρχή των τριών όχι. Πρόκειται για καλή αρχή, αλλά Πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει να την επανεξετάσουμε αν θέλουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. 36 σημεία θα ήθελα να θέσω. Τέλος πάντων, για να σοβαρευτώ, τέσσερα πολύ σύντομα σημεία. Υπόθηκε σήμερα ότι πρέπει να εντοπίσουμε την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, δύσκολη πρόκληση, αλλά για μένα οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να αφορούν τα projects, να δούμε τοπικές προκλήσεις, τοπικά ζητήματα, να τα εντοπίσουμε και να υπάρξει μια διεθνής μορφή συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων. Υπάρχει ας πούμε το Σολιτβίνο μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας. Ε, δυστυχώς η γραμμή αυτή εγκαταλείφθηκε ε, και τώρα πέφτουν μέσα στο ποτάμι πάρα πολλά άλατα τα οποία σκοτώνουν τα ψάρια και αυτό δεν είναι καθόλου καλό βέβαια. Ε, η μακροπεριφερειακή στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα και αυτή τη στιγμή ε, προσπαθεί να υπάρξει ένα έργο για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο της περιφέρειας ε, του Δούναβη. Αν είχε χρησιμοποιηθεί σωστά η στρατηγική, ενδεχομένως το πρόβλημα να μην είχε προκύψει και να μην είχε συμβεί ό,τι συνέβη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά όλα αυτά τα έργα, τα projects που μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον για την αποφυγή τέτοιου είδους περιπτώσεων. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι ακόμη νέες. Νομίζω ότι όλοι μπορούν μπορούμε να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Ε, χρειαζόμαστε περισσότερες ε, εμπειρίες ακόμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να αφήσει ακόμη το χέρι των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Χρειαζόμαστε ακόμη καθοθήγηση, υποστήριξη. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να είναι αποτελεσματικές αυτές οι στρατηγικές και δεν βλέπω ε, βάσει των εξελίξεων αυτή τη στιγμή ότι θα μπορέσει να συμβεί αυτό χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Βρυξελών γενικότερα. Ελπίζω να μην έχω εξαντλήσει τα δύο λεπτά μου. Η συνεργασία μεταξύ των μακροπεριφερειακών στρατηγικών πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί και ένας πρακτικός τρόπος για να το κάνουμε αυτό στο ετήσιο φόρουμ ε, στις 18 και 19 Οκτωβρίου το, η τελευταία ε, ε, ολομέλεια έχει αφιερωθεί στην εξέβρεση τρόπων για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας. Έχουμε καλέσει τις προεδρίες των ε, υφισταμένων μακροπεριφερειακών στρατηγικών και προσπαθούμε να αναζητήσουμε και συγκεκριμένα επόμενα βήματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τελευταία δύο λεπτά, δύο λεπτά ε, για τον τελευταίο μιλητή μας τον κύριο Φάβια. Ε, θα προσπαθήσω και εγώ να δώσω πέντε απαντήσεις στις πέντε ερωτήσεις. Ποιο ε, χρηματοδοτικό ε, πλαίσιο είναι ανθρώπινο. Το πλαίσιο, κατά την άποψή μου, η πολιτική συνοχή είναι ο λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα με τα χαράς ε, θα ήθελα διεύρυνση της πολιτικής και επίσης ε, το ανθρώπινο δηματικό το οποίο θα μπορεί να συμμετέχει στη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Ε, αναφέρθηκε εκπρόσωπη τη Επιτροπή στην ανάγκη να ενισχύσουμε τις διοικητικές δυνατότητες σε κάποιες χώρες. εν μέρη στα νέα κράτη-μέλη και στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κίνητρα ε, θα πρέπει να δώσουμε, θα πρέπει να είναι κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση, θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, είναι για να ενοποιήσουν και να ε, κάνουν πιο συνεκτική την, την ένωση, όχι να τη διαιρέσουν και ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες. Κάποιες μακροπεριφέρειες ε, μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, τη σημαία της περιφερειακής ε, ανάπτυξης, κάποιοι άλλοι της εθνικής. Πρέπει λίγο να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία και να τα βρούμε τη χρυσή τομή αναπερίπτωση. Εγώ αναφέρθηκα ήδη στην εμπειρία ε, της UCR που είναι από τη μία και της άλλης στρατηγικής που είναι από την άλλη. Είναι δύο διαφορετικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Και εγώ προτείνω ισορροπία. Αυτή είναι η απαραίτητη ανάγκη. Μπορείτε να εκχωρήσετε εξουσίες όπου θέλετε, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει ισορροπία ε, κάποια στιγμή παντού. Οι μακροφερειφερειακές στρατηγικές είναι μέσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να το χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει στρατηγικά ζητήματα. Βεβαίως, αυτή είναι η προστιθέμενη της αξία. Το βρήκατε. Βρήκατε, στοχεύσατε ακριβώ στο κέντρο. Και μάλιστα εγώ γι' αυτό σας είπα στην παρέμβασή μου ότι πρέπει να το προωθήσετε όπως μπορείτε, αλλά με διαφορετικό τρόπο για την κάθε περίπτωση. Τώρα, όπως σα είπα, η πολιτική συνοχή είναι ο λόγο ύπαρξη. Τι μπορούμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες τη διακυβέρνηση. σίγουρα τις διαδικασίες. Η διακυβέρνηση είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα μπορούσαμε να πλουστεύσουμε, αλλά οι αρχές της μακροπεριφέρειας είναι αυτές που θα βρουν την καλύτερη δυνατή διακυβέρνηση και κάποια στοιχεία θα γίνουν περιτά από μόνα τους και θα ξεπεραστούν. αν είσαι χρήσιμος, μένεις, αλλιώς ε, σε σβήνω από το χάρτη. Νομίζω ότι απάντησα στις πέντε ερωτήσεις. Κάποιος είπε από τους ομιλητές να ρωτήσουν τον κόσμο αν γνωρίζει τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Ρωτήστε λοιπόν τους ανθρώπους της περιοχής σας, ε, αυτήν που εκπροσωπείτε εσείς, ποια είναι η σωστή απάντηση. Είναι τοπική ή είναι περιφερειακή ε, ή μακροπεριφερειακή και θα πάρετε την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε και τους προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι υπάρχει η παρουσία σας εδώ στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή όμως όταν θα συζητήσουμε την έκθεση για την εφαρμογή. Σήμερα ε, ασχοληθήκαμε με την άποψη των εμπειρογνωμόνων που είχαμε καλέσει για το εργαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καθυστερήσει ως συνήθως. Και περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, προετοιμασία τη θέση του Κοινοβουλίου για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε τη γνωμοδότηση ε, τη Επιτροπή Ρέτζη, συντάκτη είναι ο κ. Ντέρεκ Βον και θα ακούσουμε την παρουσίασή του για τη γνωμοδότηση και μετά θα δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές. Η πρόταση για κατάθεση τροπολογιών τέλος ε, της ημέρας ε, Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου διότι πρέπει να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα της Μόδιας Επιτουσίας Επιτροπής Επιτροπής Προϋπολογισμών βλέπω ότι ο κύριος Όλμπρεχτ που είναι εισηγητές είναι εδώ Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Βόν έχετε το λόγο Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Θα Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γιάνν που είναι εδώ να παρακολουθήσει τη συζήτησή μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας. Ε, πολύ πρόσφατα, μάλιστα πριν από δύο εβδομάδες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας ε, για το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Και σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων αναφέρθηκα σε αυτά τα οποία θεωρώ τα ουσιαστικά ζητήματα για την Επιτροπή μας. Για παράδειγμα, αναφέρθηκα στην ανάγκη να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 και ξέρουμε ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο διότι ο προπολογισμό ε, θα είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Ε, πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση και ότι η πολιτική συνοχής θα παραμείνει το βασικό επενδυτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης ανέφερα ότι θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να βρούμε έναν τρόπο να δημοσιοποιήσουμε περισσότερο τα ωφέλη τη πολιτική συνοχή. Δυστυχώ, πιστεύω ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλοί δικαιούχοι που δεν ξέρουν καν ότι είναι δικαιούχοι. Το βλέπω και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ουαλία, αλλά το βλέπω και όταν πηγαίνουμε σε αποστολέ με την Επιτροπή Ρέτζι ή με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, στην οποία συμμετέχω επίση. Διακόπτη Πρόεδρος, ε, κυρίες και κύριοι σας παρακαλώ πολύ Εάν ε, δεν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη συζήτηση για το μέλλον των πολιτών ε, δημοσιονομικών πολιτικών, παρακαλώ μπορείτε να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε κύριε Βόν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ε, Καλό είναι να έχουμε μία συνεδρία σε εξελίξη, φαίνεται να έχουμε δύο-τρει ταυτόχρονα. Θεωρώ λοιπόν, ε, έλεγα και προηγουμένω, ότι καλό είναι να δημοσιοποιήσουμε τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το Ταμείο Συνοχή. Επίση, ε, να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια τη πολιτική συνοχή θα βασίζονται σε ενισχύσει και να μην υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή για να αυξηθεί ο αριθμό των δανείων αντί για των ενισχύσεων. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Επίση, ε, θα πρέπει να γίνει περίοδος του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου 5 ε, 5, ε, όχι 5 και αυτοί που θέλουν να διατηρήσουν 7, να έχουμε ένα μέσο όρο, δηλαδή μια κατάλληλη χρυσή τομή θα είναι το 5 5 ίσως. Ε, ε, επίσης είπα ότι θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες συνέργειες μεταξύ κονδυλίων. Αν μπορέσουμε να συνδυάσουμε διάφορα ταμεία, για παράδειγμα, θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιρροή. Και ένα από τα βασικά στοιχεία, τα οποία έφυξα και στην παρέμβασή μου τότε, ήταν αυτό. Τα έχω συμπεριλάβει όλα αυτά στο σχέδιο γνωμοδότησης, ε, τα έχουν οι συνάδελφοι, αλλά και κατά την ανταλλαγή απόψεων αρκετοί συνάδελφοι έκαναν αρκετές παρατηρήσει τις οποίες προσπάθησα να συμπεριλάβω στην πλειοψηφία τους ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης. Για παράδειγμα, έχω συμπεριλάβει την ανάγκη να ε, ε, εγκρίνουμε το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν για να υπάρχουν και κανονισμοί για την πολιτική συνοχή και να ξεκινήσει η εφαρμογή των πολιτικών συνοχή το συντομότερο δυνατόν. Κάθε φορά που έχουμε νέο πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο έχουμε καθυστερήσει και αυτό δημιουργεί και προβλήματα στην εφαρμογή και στην απορρόφηση των κονδυλίων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Επίσης ανέφερα και ε, μετά από σχόλια των συναδέλφων ότι θα πρέπει να αναφέρουμε και την πρόκληση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ συγγνώμη εκ βάθους καρδίας, ε, νιώθω ντροπή πραγματικά γι' αυτό, αλλά ε, αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις υπάρχουν 8 ποσοστίες μονάδες διαφορά μεταξύ αυτών που θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών που θέλουν να αποχωρήσουν. Συνειδητοποιεί δηλαδή ο κόσμος το ολέθριο σφάλμα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να το ανατρέψει αυτό. Τουλάχιστον όμω υπάρχει μια κίνηση προ τη σωστή κατεύθυνση. Αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα υπάρχουν τεράστιε συνέπειε φυσικά για τον προπολογισμό τη Ένωση και θα πρέπει να το αναφέρουμε στο σχέδιο γνωμοδότηση. Επίσης ανέφερα ότι οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να επικαιροποιηθούν για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε νέες προκλήσεις και στην ανταλλαγή απόψεων συζητήσαμε και κάποιες από αυτές τις προκλήσεις. Είδαμε όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν και κάποια στοιχεία τα οποία έθιξαν οι συνάδελφοι ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης τα έχω συμπεριλάβει και ε, πιστεύω ότι θα χαρούν οι συνάδελφοι γι' αυτόν. Και επειδή ε, έχουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων και έχω και το πρώτο σχέδιο γνωμοδότηση έτοιμο, έχουμε και το, σχέδιο, το έγγραφο προβληματισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και αυτό το έγγραφο προβληματισμού και να αντανακλάται και κάποιο στη γνωμοδότησή μα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να υποβάλω και κάποιε τροπολογίε ο ίδιο, ώστε να λάβουμε υπόψη και κάποια από τα στοιχεία τα οποία αναφέρει και ο Επίτροπο Προπολογισμού σε αυτό το έγγραφο προβληματισμού παράδειγμα, θεωρώ ότι θα ήταν καλό για μα να αναφέρουμε και την προστιθέμενη αξία τη πολιτική συνοχή. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι η πολιτική συνοχή όντω έχει επιρροή και είναι αποτελεσματική και αλλάζει τα πράγματα. Εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχή για το μέλλον, πρέπει να σταθούμε σε αποτελέσματα, σε επιδόσει και να δείξουμε ότι όντω έχει προστιθέμενη αξία η πολιτική συνοχή. Θέλω λοιπόν να προσθέσω αυτό. Θα ε, ήθελα επίση να πούμε, όπω λέγαμε πάντα στο παρελθόν, ότι η χρηματοδότηση τη πολιτική συνοχή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλε τι περιφέρειε. Διότι αν δούμε το έγγραφο προβληματισμού, αμφισβητείται αυτό το γεγονό εκεί. Και θα πρέπει να έχουμε εδώ πολύ στεναρή στάση. Ε, κάθε περιφέρεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει χρηματοδότηση από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχή. Και νομίζω ότι θα πρέπει, επειδή αναφέρεται στο έγγραφο προβληματισμού, να λέμε και εμεί κάτι γι' αυτό στη να πούμε και κάτι για ένα σύνολο κανόνων για όλα τα ταμεία. Το έγγραφο προβληματισμού κάνει κάποια πρόταση να έχουμε ένα ταμείο, λέει, ε, και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων επ' αυτού. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύνολο κανόνων. Ε, τώρα ένα ταμείο προσωπικά καταλαβαίνω ότι έχει κάποια ωφέλη, αλλά μπορεί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ε, μπορεί να μην θεωρούν ότι είναι και η πιο δελαστική πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων επ' αυτού. Ε, θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να πούμε και δύο λόγια για την εξάντε και την ε, δημιουργία δυνατοτήτων, το capacity building. Ε, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στο παρόν πρόγραμμα και σε πολλές περιφέρειες έχουν την αίσθηση ότι ένα από τα προβλήματα ε, της χαμηλής απορρόφησης είναι ακριβώς ε, το θέμα της εξάντερεσιμότητας και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες να δαπανηθούν τα κονδύλια. Θα πρέπει ίσως να θίξουμε και αυτό. Αυτά κατά με ήταν τα αρχικά θέματα, κάποια θέματα τα οποία συμπεριέλαβαν οι συνάδελφοι στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων, συν κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να προσθέσουμε μετά από τη δημοσίευση του εγγράφου, προ... του εγγράφου προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων επ' αυτού, αλλά και στο μέλλον βέβαια και των σχεδόν εισηγητών και ε, περιμένω και τις τροπολογίες όπως είπατε, ε, τις οποίες πρέπει να υποβάλλετε μέχρι τις 4 ε, Σεπτεμβρίου για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε με τους συναδέλφους όλα αυτά και να πω στους συναδέλφους ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι σημαντική για την Επιτροπή Ρέτζη. Μας δίνει την ευκαιρία να ε, κοινοποιήσουμε και τις απόψεις μας ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, αλλά κυρίως για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι μοναδική ευκαιρία λοιπόν να γνωστοποιήσουμε τις απόψεις μας και ε, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι αυτό θα θίξουν σήμερα και στις τροπολογίες που θα μου υποβάλουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σπυράκη και οδησηγήτρια. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι εισηγητή. Είναι πράγματι πολύ σημαντική η προετοιμασία που κάνατε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Θα ήθελα καταρχήν να θέσω το θέμα του reflection paper από την πλευρά της Κομισιόν και να πω ότι είναι ανάγκη να αντανακλάτε σε αυτή την γνωμοδότηση ο προβληματισμός που υπάρχει στο reflection paper και ιδιαίτερα τα όρια της ευελιξίας την οποία προτάσει το reflection paper. Είναι σαφές ότι ο όρος flexibility κυριαρχεί εκεί. Θα είναι λοιπόν καλύτερο εμείς ως Επιτροπή Ρέτζι να θέσουμε ακριβώς το όριο στο οποίο θα κινηθεί πρώτον η ευελιξία και δεύτερον πόσο αυτή θα αφορά ειδικά το κομμάτι των κοντιλίων συνοχής. Επίσης θα ήθελα να, να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της συμπληρωματικότητας και της προσθετικότητας των ευρωπαϊκών πόρων, δεδομένου ότι είναι προφανές ότι η νέα τάση, τάση την οποία εκτιμώ ότι δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε και καλώς δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε ζητώντας να συμβαίνει ό,τι συνέβαινε πριν από 7 χρόνια, είναι η συμπληρωματικότητα των πόρων. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα αυξήσουμε τη μόχλευση μεταξύ κονδυλίων που προέρχονται από τον προϋπολογισμό, κονδυλίων που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και κονδυλίων που προέρχονται από ανταγωνιστικά προγράμματα όπως είναι το Horizon και το SEF. Βεβαίως πρέπει σημαντικά να επιμείνουμε στην απλοποίηση και εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας ότι χρειαζόμαστε έναν κανονισμό για κάθε ταμείο και όχι ένα ταμείο για, τη για, πάσα χρήση και για πάσα νόσο. Και κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι είναι σαφές ότι η, η προστιθέμενη αξία της ε, πολιτικής συνοχής πρέπει να, να μέσα από τη δική μας νομοδότηση και αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με μια ε, μορφή επικοινωνίας η οποία θα έχει να κάνει όχι μόνο με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες αλλά με τους, με τους ε, ε, stakeholders στο έδαφος, δηλαδή με, τους, με τα πανεπιστήμια, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες που τελικά επωφελούνται από αυτή την πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή μας, ο οποίος ε, πραγματικά συμπεριέλαβε έναν μεγάλο αριθμό ε, των προτάσεών μας. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ε, αδυναμίες στο σύστημα ε, χρηματοδοτικού προγραμματισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μαζεύονται οι λογαριασμοί που δεν έχουν πληρωθεί και ε, καθυστερούμενες όφιλες από την προηγούμενη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ε, για την αρχή κάποιων προγραμμάτων ε, την ε, περίοδο 2012 με 2020 έγινε κάποια μεταφορά από την προηγούμενη περίοδο και αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην εφαρμογή της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και ελπίζουμε αυτό το πρόβλημα να μην μεταφερθεί και στην επόμενη περίοδο. Ε, θα έπρεπε λοιπόν η ολοκλήρωση ε, να, του προγραμματισμού να γίνει πριν από το τέλος του 2000, ε, πριν από το 2018 για να μπορέσει να γίνει η εφαρμογή γρήγορα και να αρχίσουμε από το 2021 να εργαζόμαστε γρήγορα και να μην χρειάζεται να έχουμε καθυστερούμενα από την προηγούμενη περίοδο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση και μια ρυθμιστική προσέγγιση της πολιτικής συνοχής, ώστε οι διάφοροι κανόνες να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό τρόπο και η χρηματοδότηση να είναι και εκείνη πιο αποτελεσματική. Η συνέχεια η ρυθμιστική θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής στο πλαίσιο της Ένωσης και γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει ένας εφαρμοστικός κανονισμός ο οποίος θα αλλάξει ε, όσο το δυνατόν λιγότερο τους κανόνες ε, για, την, ε, για, για τις για, την, για τις προμήθειες, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα συνεχίσω στα βουλγαρικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βόαν για το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ήθελα να πω ότι τον υποστηρίζω στις περισσότερες από τις τροπολογίες που υπέβαλε. Νομίζω ότι τόνισε τη σημασία της ε, πολιτικής συνοχής προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων των προκλήσεων βέβαια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, ε, τόνισε την αναγκαιότητα περισσότερης ευελιξίας για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ προκλήσεις. Πρέπει να μπορούμε τις επιδοτήσεις να τις συνδυάσουμε με τα ε, ευρωπαϊκά ε, διαρθρωτικά ε, και επενδυτικά ταμεία. Πολλά ε, προγράμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν ε, να συνδυαστούν με το ε, ΕΦΣΙ, όπως επίσης ε, και με διάφορα καινοτόμα προγράμματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας πολλαπλασιαστικός αντίκτυπος στον προϋπολογισμό. Η συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες είναι επίσης πολύ σημαντικός. Η περίοδος 5 συν 5 για την επόμενη περίοδο με βρίσκει σύμφωνη. Επίσης πιστεύω ότι το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες με μεγάλη προστιθέμενη αξία που ενισχύουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποτελεσματική ε, κατανομή των πόρων. Πρέπει να δούμε την προστιθέμενη αξία ε, των ε, επενδύσεων στο επόμενο πι και είναι επίσης πολύ σημαντική και η εδαφική συνεργασία, το πρόγραμμα, τα προγράμματα Interreg για παράδειγμα, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για τα κοινά προγράμματα, τα οποία είναι διασυνοριακά για πάνω από μία χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης προπολογισμό τη Ένωση πρέπει να συμπληρώνει τον εθνικό προπολογισμό και να εστιάζεται σε εκείνου του τομεί ε, στου οποίου ε, ο εθνικό προπολογισμό δεν είναι καλά στοχευμένο. Είναι σημαντικό το επόμενο ΠΔΠ να υποστηρίζει ολόκληρη τη διαδικασία των ευρωπαϊκών εξαμήνων και ειδικότερα τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, δημιουργώντα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον. Χρειαζόμαστε επιπλέον διαφάνεια για τι επενδύσει εντό τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύξηση της, ευαισ... της ε, ε, ευαισθητοποίησης και της ορατότητας ε, του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Και τέλος, το επόμενο πι πρέπει να εστιάζεται σε ευέλικτη χρηματοδότηση, στο συνδυασμό χρηματοδοτικών μέσων, την αστική ανάπτυξη, την εδαφική συνεργασία, την ανάπτυξη, την καινοτομία και να συνδέεται περισσότερο με την οικονομική διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Αυτή ήταν η δική μου συνεισφορά ω κοιόδου εισηγήτρια. Ο κ. Σόμερ δεν είναι εδώ. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρου του σκιώδου συζητητή τη ομάδα μας, του κυρίου Μαρζή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Οβόν, τον εισηγητή μας, για την ε, εξαιρετική προετοιμαστική δουλειά που έχει γίνει και να πω ότι συμφωνούμε με πάρα πολλέ από τις προτάσεις του όπως τις κατέθεσε και με τροπολογίες και όπως τις παρουσίασε σήμερα. Το πιο σημαντικό κατά την άποψή μας είναι να επιδιώξουμε και να επιμείνουμε η Επιτροπή Περιφερειών να παραμείνει ισχυρή η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετά το 2020. Γιατί μετά το Brexit και τις επιπτώσεις του στον προϋπολογισμό υπάρχουν κίνδυνοι και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ε, βοηθούν ορισμένα πράγματα που επεσήμανε και ο, ο κ. Βόν. Πρώτον, να προβληθούν τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών συνοχής, αλλά και να προβληθεί το τι ζημιά θα είχε γίνει αν δεν υπήρχαν οι πολιτικές συνοχής, γιατί παρά τις πολιτικές συνοχής τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μεγάλη αύξηση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Που σημαίνει ότι χωρίς πολιτικές συνοχής ή με πιο αποδυναμωμένες πολιτικές συνοχής οι ανισότητες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες εκρηκτικέ. Μια ακόμη παρατήρηση αφορά στη μορφή της αξιοποίησης των πόρων. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι αυτή πρέπει να έχει κυρίως τη μορφή των ενισχύσεων και όχι των α, δανείων μέσω της μόχλευσης. Και πιστεύω ότι το κείμενο προβληματισμού, το έγγραφο προβληματισμού που παρουσίασε η Κομισιόν εμπεριέχει ε, και ορισμένους κινδύνους για την πολιτική συνοχής, κυρίως μέσα από μια πολύ ελαστική δυνατότητα ερμηνείας του όρου ευελιξία. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Η Επίτροπος, ε, η κυρία Κρέτσου, υποστηρίζει θερμά τις πολιτικές συνοχής και γι' αυτό έχει την Επιτροπή μας σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, αλλά μέσα στην Κομισιόν υπάρχουν και ισχυροί αντίπαλοι της πολιτικής συνοχής που επιδιώκουν να την αποδυναμώσουν. Και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή η προσπάθεια αποδυνάμωσης της πολιτικής συνοχής να μην καρποφορήσει. Συμφωνώ επίσης ότι χρειάζεται απλοποίηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ένα ταμείο. Σημαίνει ένας κανονισμός, όπως ήδη υπόθηκε, για κάθε ταμείο. Αλλά το ένα ταμείο έχει κινδύνους. Και επίσης πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την περίοδο 5 συν 5 με σαφήνεια, όπως ήδη υπόθηκε από τον κύριο Βόν. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Ομαρζή, ε, και με τις τροπολογίες που θα καταθέσει εκ μέρους της ομάδας, σε στενή συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους κοιόδη εισηγητές των πολιτικών ομάδων, θα συμβάλλει έτσι ώστε η opinion εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειών να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή και υποστηρικτική για τη συνέχιση των πολιτικών συνοχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόπιος και ο συζητητής. Ε, Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι η πολιτική συνοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Η γνωμοδότηση πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Ο εισηγητής ε, έλαβε υπόψη του όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν και αν έχουμε αρνητικές επιπτώσεις από το Brexit, προφανώς και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην πολιτική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να αποδείξουμε σε συναδέλφους από άλλες επιτροπές, αλλά και στην ευρωπαϊκή πολιτική, ότι η πολιτική συνοχή ε, δεν είναι λιγότερο σημαντική από άλλες πολιτικές. Ίσως μπορεί κανένα να θεωρεί ότι η πολιτική συνοχή είναι μια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Μπορεί. Υπάρχουν ε, διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής και θα ήταν καλό αν τα κονδύλια που ανήκουν σε στην πολιτική συνοχή μέχρι και 30% να πήγαν σε όλες ε, τις περιφέρειες ανεξάρτητα από την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οι διάφορες περιφέρειες ή αν θέλετε ορισμένες περιφέρειες δεν παίρνουν καθόλου χρήματα, καμία χρηματοδότηση. Παραδείγματο χάρη υπάρχει το εργαλείο Leader Plus, το οποίο ισχύει για όλες τις ε, περιφέρειες. Και νομίζω ότι Θα πρέπει να υπάρχει όμως ε, χρηματοδότηση και για περιφέρειες που μέχρι τώρα δεν είχαν καμία χρηματοδότηση. πολιτική επενδύσεων και αυτή είναι πολύ σημαντική. Γιατί στη δική μου την περιοχή, στη Βαλτική, ανέρχεται στο περίπου 10%. Και ακόμα δεν προβλέπονται χρήματα για την περίοδο μέχρι το 2020. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτά τα κενά, δημιουργείται μια μεγαλύτερη καθυστέρηση που οδηγεί σε δάνεια και αυτά μετακυλίονται σε άλλες επόμενες περίοδους. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται προβλήματα και νομίζω ότι πρέπει αυτήν την αρχή να την διαφυλάξουμε καλύτερα. Για το πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο είχαμε το σενάριο πριν από δύο εβδομάδες. Μας τα παρουσίασαν η Επίτροπος Κρέτσου και ο Επίτροπος Έτιγκερ για το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθόλου ρόδινο δεν φαίνεται για την πολιτική συνοχή. Η γνωμοδότηση του συναδέλφου Βον έχει κάποιες ε, πολιτικές θέσεις οι οποίες με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Για παράδειγμα, πρέπει να βρούμε μια γρήγορη συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις και συνεπώς να διαπραγματευτούμε για την πολιτική συνοχή στο συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να υπάρξει επαρκής προϋπολογισμός ε, για να γίνουν επενδύσεις για τους πολίτες, ε, για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τους πολίτες. Επίσης, κάποιες ενισχύσει που λέει ο συνάδελφο ότι θα πρέπει να δίνονται μόνο σε κάποιε περιπτώσει. Εγώ επιμένω εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει προστιθόμενο αξία και ε, χαμηλό ε, συντελεστή κινδύλου. Επίση, συμφωνώ για την προτίμηση ενό πι 5 συν 5 ετών, αλλά και σε αυτή την περίπτωση με μία διευκρίνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβλέψουμε αναθεώρηση, ενδιάμεση αναθεώρηση, ε, στο τέλο των ετών. Ε, όπως είδαμε αυτούς τους μήνες, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ε, του θέματος για τις φυσικές καταστροφές, ε, πρέπει η πολιτική συνοχή να γίνει πιο αξιόπιστη και να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία. Και θεωρώ ότι η ε, μετανάστευση και τα θέματα ασφάλειας ε, ε, και προστασίας θα πρέπει να εξετάζονται με διαφορετικό τρόπο από την πολιτική συνοχή. Επίσης πρέπει να βρούμε μια σύντομη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και να πριτανεύσει κοινή λογική και από τις δύο σκοπιές. Δεν μπορούν οι πολίτες να περιμένουν για να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εγκριθεί τελευταία στιγμή. Ε, πρέπει να έχουμε μια καλύτερη πολιτική συνοχή, να γίνει πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πραγματικά να ε, αφορά την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Να ελέγχουμε ποια προγράμματα στη συνέχεια εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος ε, για να υπάρχει μια ισορροπία. Ισορροπία μεταξύ της απλοποίησης των διαδικασιών και ταυτόχρονα του ελέγχου για την ποσότητα αλλά και την ποιότητα της δαπάνης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχω κατάλογο των υπολείπων ομιλητών. Ο κύριος Βαρκάρθερ Σίσο έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και κάποιους μήνες ασχολούμαστε ε, και εμβαθύνουμε περισσότερο στα θέματα που αφορούν την πολιτική συνοχής. Και γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2020 και μετά, ουσιαστικά θεωρούμε δεδομένο ότι κατά πάσα πιθανότητα η απαχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα προκαλέσει σεισμό στον προπολογισμό, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός χορηγός. Και φυσικά εδώ ε, έχουμε πάρα πολλά τα οποία διακυβεύονται στις διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και πρέπει να τις παρακολουθούμε πάρα πολύ ε, στενά. Το Brexit όμως δεν είναι η μόνη υπόθεση ε, που θα απασχολήσει τη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Υπάρχει όλη η συζήτηση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Πολιτικού Δημοσιονομικού Πλαισίου που πάλι η πολιτική συνοχή είναι στοιχείο κλειδί οι νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση θα πρέπει ε, να λαμβάνουν υπόψη τους και την ευρωπαϊκή διάσταση της συνοχής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα ε, θετικά στοιχεία για να προωθήσουμε τη συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Ενισχύσεις, δάνεια, χρηματοοικονομικά μέσα, ίσως κάποιος συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων με καλύτερη θεματική εστίαση. Όλα αυτά τα θέματα είναι ανοιχτά και υποσυζήτηση και αυτό το οποίο με ανησυχά κυρίως είναι ότι υπάρχει η πρόκληση ε, να ε, ε, απαντήσουμε με επιχειρήματα ποια είναι η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής. Πρέπει λοιπόν να παρουσιάσουμε απτά αποτελέσματα, ώστε κανείς να μην μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να θεωρούμε την πολιτική συνοχή το βασικό στοιχείο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ολοκληρώνω με το εξή, θα πρέπει να προχωρήσουμε την απλοποίηση. Τη ζητάμε συνεχώ ε, στην Επιτροπή μα στη διάρκεια όλη αυτή τη θητεία και σίγουρα η πρόταση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο ε, θα πρέπει να αντανακλά και κάποια πρόοδο προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Βαν Μίλτεμπεργκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την πρόεδρό μας. Εγώ θα συνεχίσω στα αγγλικά Καταρχά θα ήθελα να πω ότι η παρατήρηση έχει ήδη γίνει ότι η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής, ε, ε, η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ή άλλως θα αναστατωθεί γιατί όταν μιλάμε για το ίντερνετ και πολύ σωστά το είπατε κι εσείς ε, κυρία Πρόεδρε είναι ένα πρόγραμμα του οποίου ο προπολογισμό πρέπει να αυξηθεί. Όμω το Brexit θα έχει ήδη έναν αντίκτυπο στη διασυνοριακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για την διακρατική ε, συνεργασία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε αυτάπάτε, ε, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια λογική πολιτική, μια περιφερειακή πολιτική, συγγνώμη, που μπορεί να παραμείνει όπω σήμερα. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για να υπάρχει υπάρχει μια περιφερειακή πολιτική, ε, μια δεύτερη εκδοχή ε, για να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε, να την εξελίξουμε με καλύτερο τρόπο, να επικεντρωθούμε περισσότερο στις επιδόσεις, στα αποτελέσματα και στις πραγματικές ανάγκες ε, ε, και τον τρόπο χρηματοδότησής της ε, από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Δεύτερο σημείο, ο συνδυασμός των ε, καινοτόμων και χρηματοδοτικών μέσων. Νομίζω ότι η παράγραφος 3 είναι λίγο αμυντική ε, όσον αφορά ε, το ΕΦΣΙ, ούτως ή άλλως το ΕΦΣΙ τρίτη ε, εκδοχή μπορεί ούτως ή άλλως να συνδυαστεί και να επιφέρει νέες επενδύσεις στην Ευρώπη. Όσον αφορά το 5 5 και την προγραμματική περίοδο, τίθεται το ερώτημα πότε πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση όμως. Τώρα έχουμε μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Πρέπει να γίνεται κάθε δυόμιση χρόνια, δεδομένου ότι κάθε φορά έχουμε μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση αλλά μερικέ φορέ δεν υπάρχει αρκετό περιεχόμενο για να γίνει μια πραγματική ειδική αξιολόγηση που να μα επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα από τι προηγούμενε περιόδου. Πρέπει να το κάνουμε λοιπόν κάθε δυόμιση χρόνια ή κάθε πέντε χρόνια, ε, το οποίο επίση είναι μια δυνατότητα. Συμφωνώ με τι παρατηρήσει σα, κύριε εισηγητά ότι η περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να καλύπτει όλε τι περιφέρειες Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπάρχουν πολλές ανάγκες, ε, ακόμη και στις πολύ ανεπτυγμένες περιφέρειες χρειάζεται η ενίσχυση της ε, καινοτομίας, της ανάπτυξης ε, και της έρευνας και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν συζητήσαμε τους θεμέλιους λήθους της πολιτικής συνοχής ε, αναφερθήκαμε στην κάλυψη όλων των, περιφερειών της Ένωσης και η τελευταία μου παρατήρηση που είναι περισσότερο μία σκέψη όταν μιλάμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μήπως θα μπορούσαμε να αρχίσουμε και τη συζήτηση για τα ε, κονδύλια που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίηση και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ε, με το, γραφείο, με το ε, ταμείο αυτό και στο πλαίσιο των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα. Ε, καταλαβαίνω βέβαια ότι πρέπει να διαλέξουμε τις μάχες που θα δώσουμε και να κάνουμε την περιφερειακή μας πολιτική πάλι πολύ σημαντική και πολύ μεγάλη μετά το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Μπρέσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν επιτρέψτε μου και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την πολύ καλή δουλειά που κάνει με κέφι, με πάθος η δουλειά που έχει σχέση με θέματα προϋπολογισμού. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις. Αν διαβάσουμε προσεκτικά την τρίτο άρθρα 3.10 και 3.11 των συνθήκων, εκεί που γίνεται λόγος ε, για τις ε, χρηματοδοτικές ε, διατάξεις, θα διαπιστώσουμε ότι το οδηγό νήμα των συνθήκων, οποτεδήποτε πρόκειται για νέε λειτουργίε, αρμοδιότητε και πολιτικές, χρειάζονται και νέοι πόροι. Αυτά λένε οι συνθήκε. Ενώ στη συζήτηση εστιάζουμε την προσοχή μας στο πώ θα αφαιρέσουμε κονδύλια από πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτές είναι δύο. Δύο είναι αυτέ. Είναι η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχή. Πώ θα αφαιρέσουμε από εκεί κονδύλια για να κάνουμε κάτι άλλο και ενδεχομένω ε, και για να καλύψουμε κάποιο κενό που θα προκύψει ενδεχομένω από την ε, αποχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι σωστό. Το έγγραφο για τους ιδίους σπόρους και η σχετική μελέτη που παρουσιάστηκε για τους ίδιους σπόρους, εκεί αναφέρεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν ήδη πόροι για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι επιβαρύνοντας πολίτες, αλλά χρησιμοποιώντας τα εργαλεία εκείνα που επιτρέπουν τον έλεγχο της παγκοσμιοποίησης. Το λέω έτσι πολύ συνοπτικά, αλλά ξέρετε ακριβώς τι είναι. Ως εκ τούτου προς τα εκεί πρέπει να πιέσουμε και να ζητήσουμε οι παραδοσιακοί πόροι, τα κονδύλια αυτά να παραμείνουν στην πολιτική της συνοχής. Γιατί είδαμε στο τελευταίο φόρουμ ότι η πολιτική συνοχής ε, αρχίζει να παίζει τον πραγματικό της ρόλο. Αυτή η σκληρή οικονομική κρίση δεν μπορούσε δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με την πολιτική συνοχή. Ε, χρειαζόντουσαν και άλλα εργαλεία πέρα από αυτή την πολιτική συνοχή. συνοχής. Όμως η πολιτική συνοχής τη στιγμή που βγαίνει κανείς από την κρίση έρχεται πλέον ο ρόλος της, ο δικός της, ο μικροοικονομικός, δηλαδή να μειωθούν οι διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά στη σύγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ε, πολιτική συνοχή, όπως σας είπα, έχει βασικά αυτό το στόχο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι οφείλουμε να ζητήσουμε αμετάκλητα και αποφασιστικά από το Συμβούλιο να αποφασίσει ταχύτατα επί ενός θέματος. Κατά πόσον η πολιτική συνοχή θα παραμείνει μια πολιτική για όλες τις περιφέρειες. Και αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να, ε, στον μελλοντικό κανονισμό ο μελλοντικό κανονισμό να είναι προαπαιτούμενο παράλληλα με τη δουλειά που γίνεται με το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί αλλιώ, αν δεν γίνει αυτό, και σα ζητώ και συγγνώμη γιατί χτυπάει το κινητό μου, με συγχωρείτε πολύ, διακόπτει ομιλήτρια. Ε, κατά τα άλλα, ε, θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κατορθώσουμε σε αυτή τη θητεία να εγκρίνουμε μια νέα πολιτική συνοχή. Και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι όταν θα έχουμε φτάσει στην προεκλογική περίοδο θα χάσουμε τρία χρόνια για την πολιτική συνοχή. Άρα θα υπάρξει αυτόματα μείωση κονδυλίων γιατί θα έχουν περάσει κάποια χρόνια στην επόμενη θητεία χωρίς πολιτική συνοχή, γιατί δεν θα έχει εγκριθεί ο κανονισμός. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι τα δύο αυτά πράγματα να βαδίζουν εκ παραλίλου. Να ζητήσουμε το Συμβούλιο να αποφανθεί ότι πράγματι η πολιτική συνοχή πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για όλες τις ε, περιφέρειες και βεβαίως παράλληλα συνεχίζει και το θέμα του κανισμού, Γιατί ε, αν τελικά αποκλειστούν οι, οι περιοχές που έχουν σχέση με τον αγωνισμό είναι σαφές και δεν θα μπορείς να ξεκινήσει δουλειά για τον επόμενο κανισμό. Και ειλικρινά κινδυνεύουμε σε αυτή τη θητεία να χάσουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σχανίστελ Ρόε. Uh, is, is... Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η θέση του Derek Vaughan. Μας δίνει την άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου και μας δίνει και τη δυνατότητα να δούμε ότι η υποστήριξη για το Brexit μειώνεται όλο και, ε, όλο και μειώνεται. Υπάρχει ένα νέο σλόγαν. Exit from Brexit. Έξοδος από το Brexit. Αυτό νομίζω ότι έχει αντίκτυπο στο δικό μας έγγραφο και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να στείλουμε ένα πάρα πολύ ε, σημαντικό μήνυμα για αυτά τα building blocks που αναφέρονται ήδη στην έκθεση Festival να επιμείνουμε ότι πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία και ότι ο καλύτερο τρόπο να το επιτύχουμε αυτό είναι ο δικό μα τομέα. Η απλούστευση δεν είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει μόνο στα λόγια. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, όλε τι δυνατότητε που έχουμε για να ε, το επιτύχουμε, για να την επιτύχουμε και νομίζω ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες στη διάθεσή μας. Αυτό το έγγραφο ε, συζήτησης θα πρέπει να μας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσουμε σελίδα και να ε, ξεφύγουμε από λάθη του παρελθόντος. Πρέπει να καλύπτουμε όλες τις περιφέρειες και βεβαίως πρέπει να υπάρχει και κάποια αντιστάθμιση για τις ε, μειονεκτούσες περιοχές. Πρέπει επίσης να βασιζόμαστε και στην οικονομία της γνώσης. Θέλουμε να περάσουμε σε ε, συγχρηματοδότηση άνω των 60 δισεκατομμυρίων, αλλά λίγα λέγονται γι' αυτό όταν πρόκειται για την αναθεώρηση και τον ανασχηματισμό του ορίζοντα 2020. Αυτό είναι σημαντικό στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στη γνώση. Πρέπει να φέρουμε την αλλαγή και δεν έχουμε και χρόνο στη διάθεσή μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερούμε. Ο πραγματικό κίνδυνο είναι ότι αν αρχίσουμε να έχουμε ένα ενιαίο ταμείο και το συζητούμε αυτό ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα καθυστερήσουμε. Πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι γρήγορη σε σχέση με το και πρέπει επίση ε, τον συντελεστή χρηματοδότηση να τον δούμε αν έχουμε λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μας, πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση, το, το πώς τα διανύμουμε και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό. Εγώ προσφάτως εκπροσώπησα την Επιτροπή μας ε, στο άτυπο συμβούλιο και στη συνάντηση στη Μάλτα. Άκουσα τα κράτη-μέλη ε, να λένε πολύ παρόμοια πράγματα με αυτά που, λέγω, που λέγονται εδώ σήμερα ότι με το συνδυασμό διαφόρων ε, πολιτικών και διαφόρων εργαλείων μπορούμε να επιφέρουμε καλύτερη χρηματοδότηση. Και το άκουσα αυτό από τη Σλοβενία, από την Κροατία, από διάφορα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη που προσυπέγραψαν την αλλαγή της πολιτικής συνοχής δεν ε, αναφέρθηκαν ε, μόνο στις επενδύσεις. Ε, πρέπει να μπορέσουμε ουσιαστικές αλλαγές να κάνουμε στον τρόπο με τον οποίο οι περιφέρειες και οι πολίτες αντιδρούν. Πρέπει συνεπώς να τονίσουμε το ρόλο των κρατών μελών προφανώς είμαστε υπέρ του ρόλου των περιφερειών, όμως και τα κράτη-μέλη έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν όταν πρόκειται για την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης. Έχουμε επίσης μία επταετή συμφωνία με τα κράτη-μέλη και αυτό πρέπει να αποτελεί μία δέσμευση. ενισχυμένο ρόλο λοιπόν για τα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο ούτω ή άλλω πρέπει να αποτελέσει τμήμα των συνομιλιών μας με το Συμβούλιο και πιστεύω ότι υπάρχει θέληση να συνεχίσουμε να ε, επιμένουμε στην ευρύτερη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαφώς θα υποβάλουμε τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση. Όμω πρέπει να είναι σαφέ ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Ε, έχουμε και ένα ψήφισμα για την Ολομέλεια για την ευελιξία. Σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, μάλλον για την Ολομέλεια του Οκτωβρίου ε, θα είναι έτοιμο. Πρέπει αυτό να έχει το ίδιο πνεύμα με αυτό που συζητούμε σήμερα. Σε έξι μήνες ή σε ένα χρόνο θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο κανονισμό. Και νομίζω ότι αυτό θα ε, συνεισφέρει και αυτό ε, στην ε, συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Κύριε Σόλμπριχτ, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η δουλειά του Ντέρεκ ε, και το γεγονός ότι συμπεριέλαβε κάποια στοιχεία μετά από το, στο έγγραφο ε, προβληματισμού. Όμως νομίζω δύο στοιχεία υπάρχουν. Υπάρχει το μέλλον της πολιτικής συνοχής το οποίο θα συζητηθεί σε πολλά έγγραφα κατά τους επερχόμενους μήνες και το δεύτερο στοιχείο είναι η πολιτική συνοχή στο πλαίσιο του ΠΔΠ. Ε, το πρώτο ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο, το δεύτερο είναι κάπως περιορισμένο και αφορά περισσότερο τις αρχές. Το θέμα των αρχών, της πολιτικής συνοχής, ε, στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το βασικό ζήτημα, το πραγματικό ζήτημα είναι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε το ψήφισμα της Επιτροπής Προπολογισμών ε, που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Οπότε νομίζω ότι τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης προφανώς θα υποβάλουν τροπολογίες. Στο ψήφισμα θα ψηφίζουμε το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή Προπολογισμών και μετά τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Θα είναι μια αντίδραση στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής που είναι μια πολιτική δήλωση. Γιατί είναι πολιτική δήλωση, γιατί τα ζητήματα Τη επιτροπή ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η εξή. Εμείς θέλουμε να ε, δουλέψουμε εντό του πλαισίου προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τα πέντε σενάρια, στα τέσσερα εκ των οποίων η πολιτική συνοχής περικόπτεται, σε μία μόνο, ε, μόνο ένα σενάριο παραμένει ανοιχτό ή θέλουμε παράλληλα να εργαστούμε με αυτά τα ε, σενάρια, όπως είπε η κυρία Μπρέσο, να ε, θέσουμε επιτάπητο στα στοιχεία της πολιτικής ε, συνοχής και να μην συζητήσουμε ένα από τα πέντε σενάρια, γνωρίζοντας όμως τους περιορισμούς, να μιλήσουμε για την μελλοντική πολιτική συνοχής, για να το κάνω απλούστερο. Το ζήτημα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο είναι θέλουμε να μιλήσουμε για το πόσα χρήματα θα έχουμε και μετά να δημιουργήσουμε μια πολιτική ή θέλουμε να έχουμε πολιτική και μετά να συζητήσουμε τα χρήματα που θα έχουμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Γιατί να αρχίσουμε να συζητούμε τα χρήματα θα μας πούν θα υπάρχουν, μικρότερα, ε, θα υπάρχουν λιγότερα χρήματα, οπότε η συζήτηση είναι πώς θα γίνει περικοπή της ε, πολιτικής συνοχής και όχι πώς θα αναπτυχθεί. Αν συζητήσουμε την πολιτική συνοχή και το μέλλον της, ε, βεβαίως θα υπάρχουν κάποιες οικονομικές συνέπειες. Να σας πω την αλήθεια, πολύ καλή λύση δεν υπάρχει. Αλλά θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι πρώτον θα γίνει η δήλωση για την κατάσταση της Ένωσης από τον ε, ε, πρόεδρο Γιούνκερ το Σεπτέμβριο. Σαφώς θα υπάρξουν κάποια στοιχεία πολιτικής συνοχής το Σεπτέμβριο αυτό. Τον Οκτώβριο εμείς θα ψηφίσουμε το ψήφισμα στην Ολομέλεια για το έγγραφο προβληματισμού για τη μελλοντική χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε με ε, τους διαμορφωτές γνώμης από τις διάφορες επιτροπές για μια ε, έκθεση πρωτοβουλίας Επιτροπής Προϋπολογισμών με τη συμμετοχή όλων των επιτροπών που θα ψηφιστεί το Μάρτιο. Το Μάρτιο. Και μετά θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια νομοθετική πρόταση το Μάιο, Μάιο-Ιούνιο και τότε θα είναι η πραγματική αρχή μιας πολύ δύσκολης συζήτησης που θα είναι και πολύ σύντομη. Έξι-επτά μήνες. Νομίζω λοιπόν ότι όλα πρέπει να είναι έτοιμα ω τότε. Απλώς θα ήθελα να πω ότι ε, πρέπει να συνεργαστούμε στη επίπεδα διαφόρων ε, επιτροπών. Αυτή η δύσκολη πολιτική επιλογή του αν μιλάμε για πολιτική, για χρήματα ή πότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε είναι κάτι που πρέπει να ε, αποφασιστεί ή τουλάχιστον να γίνουν προτάσεις. Αλλιώς θα χαθούμε στις λεπτομέρειες και δεν είναι η στιγμή να γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να διακόψω λίγο τη συζήτηση για να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Βαρκάρθελ Σίσο. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ με τη συζήτηση από την αρχή από σήμερα το πρωί. Ξεκίνησαν καθυστερήσεις. Αν μπορείτε θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο το απογευματινό πρόγραμμα και να συζητήσουμε τη γνωμοδότησή σας το απόγευμα από τις 5 παρατέταρτο και μετά. Μπορείτε κύριε Βαρκάρσερ, ναι καταφετικά κύριε Βαρκάρσερ. Παρακαλώ. Γιατί έχουμε καθυστερήσει τώρα και ο κύριος Βαρκάρσερ ίσω πρέπει να φύγει. Ε, από πλευρά μου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο. Εάν οι υπόλοιποι συνάδελφοι θεωρούν ότι μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή, πολύ ευχαρίστω. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ στις 2.30 έχω ε, μία ανηλυμένη υποχρέωση. Ε, την έχουν οργανώσει διάφορες ε, ισπανικές αντιπροσωπείες και δεν μπορώ να απουσιάσω, είναι στις 2.30. Επομένως ε, η, η λύση ήταν να παρέμβω τώρα, αλλά δεν θα μπορούσα να παραμείνω για τη συζήτηση και αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι τι να πω εγώ, ε, τα ξέρω αυτά που θα πω. Το θέμα είναι τι θα πείτε εσείς για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε και τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και τους συναδέλφους που κάνουμε αυτή την αλλαγή για να συνεχίσουμε στις 5 παρατέταρτο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε και τη συνεδρίαση, αλλά ο κύριος Βαρκάθε, ίσως δεν μπορεί να μείνει ούτως ή άλλως να ακούσει τι θα πούν οι συνάδελφοι. Επομένως, Ίσως η καλύτερη λύση είναι αυτή. 5 ε, παρατέταρτο, το η γνωμοδότηση του κ. Βαρκάρθερ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα τη συζήτηση. Έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια. Κύριε Μάνσκουρ, ζητήσατε το λόγο, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομος, διότι σας δίνει το λόγο κατεξήρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Εδώ και δυόμιση χρόνια βρίσκομαι εδώ, σε αυτό τον Νίκο, και ακούω πολλές φορές να υψώνονται οι τόνοι για κάποιους οι οποίοι λένε ότι θέλουν να αμφισβητήσουν την πολιτική συνοχή, κυρίως το Ταμείο Συνοχής. Δεν θα ήθελα σήμερα το Brexit να αποτελέσει πρόσχημα για να αμφισβητήσουμε αυτή την πολιτική συνοχής, ακόμα και αν όντως ε, μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα είχαμε να προσάψουμε στην πολιτική συνοχής. Ε, σίγουρα υπάρχουν ε, ελλείψεις, αλλά είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει και πάρα πολλά. Έχουν επιτρέψει και σε χώρες από τις οποίες προέρχομαι και εγώ, νησιωτικές περιοχές, να μπορέσουν να έχουν κάποιες υποδομές. Και επειδή πέρασε και η ώρα, να πω το εξή. Ε, αν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που έχουμε κατά νου ε, δεν είναι ε, να προσπαθήσουμε να βρούμε χρήματα, να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλά, να σταθούμε στα πόδια μας. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Επομένω, δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να αμφισβητούμε την πολιτική συνοχή. Ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίε, θα πρέπει να παραμείνει η πολιτική συνοχή για να μπορέσει να αναπτυχθεί η πολιτική ε, και να μπορέσει να βοηθήσει και του λαού μα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ κύριε Γκίλαντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συζήτηση για την περίοδο μετά το 2020 και αν μου επιτρέπετε να συγχαρώ γενικά την Επιτροπή για την συνεπή στάση της συνέπεια λοιπόν ε, και αυτό υπάρχει ως ε, άποψη που εξάγουμε και από άλλες εκθέσεις. Έχω μόνο μία μικρή παρατήρηση που θέλω να κάνω. Αυτό που λέγεται στην αρχή, ότι θα βοηθούσε την Επιτροπή εάν κάποια στοιχεία τα οποία εντοπίστηκαν στο έγγραφο προβληματισμού ε, κατά πόσο αυτά ε, θα μπορούσαν να συζητηθούν περισσότερο ή όχι. Όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε, ο στόχος του εγγράφου προβληματισμού είναι να προκαλέσει συζητήσεις, δεν είναι να προσφέρει συγκεκριμένες απαντήσεις. Όμως ε, θέλω να υπογραμμίσω ότι εμείς ε, είμαστε υπέρ της ε, διαφάνειας, της επικοινωνίας, σημασία της ευελιξίας και επίσης είμαστε και υπέρ της ριζικής απλούστευσης. Το ριζική το λέω συνειδητά ως επίθετο το χρησιμοποιώ πριν από την απλούστευση. Η πρόκληση είναι πώς μπορεί κανείς να είναι ε, ριζικός αλλά να διασφαλίσετε και η συνέχεια των κανόνων. Δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητεί αυτές τις αρχές. Η δυσκολία είναι όπως πάντα να μεταφραστούν αυτά σε ε, κείμενο, σε νομοθετικό κείμενο. Ε, εμείς, εν πάση περιπτώσει, προσβλέπουμε στο να συνεργαστούμε με τα μέλη της Επιτροπής από αυτών των θεμάτων. Ο συγητής. Νομίζω ότι ε, υπήρχε συνένεση σε αυτή τη συζήτηση ανάμεσα στους ε, συναδέλφους ε, αλλά και με την Επιτροπή. Όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να προκύψει θέμενη αξία. Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να διατηρηθεί το υπόδειγμα των δανειοδοτήσεων, Ίσως λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και το έψι στις συνέργειες. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση ότι όλες οι περιφέρειες χρειάζονται κάποια περιφερειακά κονδύλια. Και ε, θα ήθελα να πω αυτό που ε, προβάλλω και εγώ στην έκθεσή μου να υπάρχει η διαφάνεια, οι δικαιούχοι να γνωρίζουν ότι είναι πραγματικά δικαιούχοι, γιατί πολύ συχνά αυτό δεν συμβαίνει. Συνένεση λοιπόν και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρουν τη σημασία της ευελιξίας. Το αναφέρω και εγώ αυτό στο σχέδιο της έκθεσής μου. Νομίζω όλοι θέλουμε να ε, διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αρκετή ευελιξία όσον αφορά στα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Για μένα αυτό που είναι προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να είμαστε και λιγάκι προσεκτικοί όσον αφορά την ευελιξία. Γιατί αυτό που δεν θέλουμε είναι να χρησιμοποιηθούν ε, τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για άλλους σκοπούς. Και είχαμε τέτοιου είδους περιπτώσεις στο παρελθόν. Ευελιξία ναι, αλλά να είμαστε και λιγάκι προσεκτικοί ε, όσον αφορά την ευελιξία στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το άλλο θέμα, ε, το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, κατά πόσον θα πρέπει να ισχύει εδώ το 5 συν 5 τέθηκε το θέμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Νομίζω ότι θα πρέπει μετά από πέντε χρόνια να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι ακριβώς έγινε τα πρώτα πέντε χρόνια. Θα πρέπει να λέμε ότι μετά από πέντε χρόνια δεν θα πρέπει να είναι ενδιάμεση αναθεώρηση με την του review αλλά και revision, επανεξέταση. Ε, ίσως λοιπόν θα πρέπει να είμαστε απόλυτα κατηγορηματικοί ότι θέλουμε τα πράγματα να επανεξεταστούν εκ βάθρων και όχι απλά να ε, παίζουμε παιχνίδια. Για το ένα και μόνο ταμείο φαίνεται να ε, επικρατεί άποψη ότι να υπάρχει ένας κανόνας για όλα τα ταμεία, αντί να υπάρχει ένα και μόνο ταμείο. Όπως σας είπα, μόνο δύο-τρεις άνθρωποι το έδειξαν αυτό και ακριβώς αυτό είπαν ε, στις ε, παρεμβάσεις τους. Ε, χαίρομαι σχετικά με τα πέντε σενάρια στο έγγραφο προβληματισμού Τα τέσσερα εξ αυτών έχουν σχέση με την πολιτική συνοχής και το δίλημα είναι αν θα είναι πρώτη η χρηματοδότηση ή πρώτα η πρωτη η Αυτό είναι μεγάλο δίλημα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Αλλά όπως είπε και ο Γιάν, τον Οκτώβρη θα έχουμε ένα ευρύτερο ψήφισμα ε, που θα ακολουθεί και ε, έκθεση πρωτοβουλίας. Εκεί λοιπόν ίσως μπορούμε να λύσουμε κάποια θέματα. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση. Υπάρχουν πολλά επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ε, πώς θα ήταν η ευρωπαϊκή πολιτική αν δεν υπήρχε συνοχή. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για την πολιτική συνοχής. Ε, ευσύνοπτη πρέπει να είναι η έκθεση. Δεν έχουμε πολύ χώρο, αλλά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Μπορούμε ε, να συμπεριλάβουμε στην έκθεση πολλά στοιχεία και όπως σας είπα και στην αρχή, νομίζω ότι μπορούμε να προβάλλουμε μια ουσιαστική άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι 4 Σεπτεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάσταση πολιγιών. Και το τελευταίο που θέλω να πω, κυρία Μπρέσο, μου είπαν ότι έχετε γενέθλια. Σχαρητήρια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πολύ ωραία. Λύει τη συνεδρίαση.